Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places, please, we can uh, begin with point 10 on the exchange of views with the European. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας και να κάνουμε την συζήτηση με την ε, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ε, κάπου στο κείμενο λέει ombudswoman, κάπου λέει ombudsman. Θα κάνουμε πολύ μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση αν μπούμε στο θέμα αυτό. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει. Βασικά το θέμα είναι ότι έχουμε έναν πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ καλό άτομο στη θέση του διαμεσολαβητού. Έχουμε δουλέψει συχνά μαζί τη και νομίζω ότι είναι και καλή η χρονική στιγμή για να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Κυρίως σε σχέση με θέματα διαφάνειας, εγγράφων, αλλά μην περιοριστείτε σε αυτό. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε γενικώ. Βεβαίω υπάρχουν και κάποιοι τομεί κλειδιά που σα απασχολούν. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν θερμότατα και κυρία Οράιλη, παρακαλώ έχετε το λόγο. Θα σας δώσουμε 10 λεπτά και μετά θα κάνουμε την συζήτηση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να μιλήσω σας σήμερα και να σας δώσω κάποια στοιχεία για τη δουλειά που κάνει η υπηρεσία μας ε, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν γιατί υπάρχουν κάποια θέματα κοινά. Η πολύ τραγική κατάσταση των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ε, ε, ε, ομάδα σας και έχουν έρθει πάρα πολλά αιτήματα και ερωτήσεις στην υπηρεσία μας. Βεβαίω είναι πολιτικέ συζητήσει που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τι αποφάσει των κρατών μελών που καθορίζουν πώ διαχειριζόμαστε το θέμα αυτό. Αλλά εμεί στο γραφείο μου προσπαθούμε να συμβάλλουμε κάθε φορά που μπορούμε. Όπως έχω ξαναπεί, ε, καλωσορίζω βεβαίως την ε, ε, στήριξη που δίνει το Κοινοβούλιο στην έκθεση για τον μηχανισμό συμμόρφωσης. Η πρόταση αυτή έχει γίνει δεχτή από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αυτοφυλακής και συνεργαζόμαστε στενά με την υπηρεσία έτσι ώστε ο μηχανισμός να δουλεύει όσο το δυνατόν καλύτερα. Επίσης έχω κάνει κάποιες συστάσεις στη Frontex για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαμβάνουν ε, κάποια ε, σωστή μεταχείριση όταν φτάνουν στην χώρα τους από κοινού με τις διαδικασίες που έχουν για τις επιστροφές στα κράτη-μέλη. Οι επιχειρήσει επίση υποχρεωτική επιστροφή ε, από τα κράτη-μέλη ε, ε, εμπίπτουν σε ένα πλαίσιο γενικών δραστηριοτήτων και βεβαίω θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το τι γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε επιτυχώ σε άλλο ένα ερώτημα στην Frontex για την πρόσβαση στα έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049 που έγινε από έναν δημοσιογράφο που έψαχνε κάποιες εκθέσεις για σοβαρά κρούσματα σε επιχειρήσεις της Frontex στη Βουλγαρία. Μετά το ερώτημα αυτό έγινε η έρευνα των, ε, των, ε, των εγγράφων και βρέθηκε η λύση. Τα έγγραφα δηλαδή δόθηκαν στην δημοσιότητα και έκλεισε η έρευνα επιτυχώς. Και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τη Frontex για, την πολύ, για το πνεύμα συνεργασίας που δείχνουν. Συνάδελφοι, ξέρω ότι η Επιτροπή αυτή είναι πραγματικά ιδιαίτερο συνεργή στο θέμα του Brexit. Έχουμε λάβει 7 ε, ε, παράπονα για, που σχετίζονται με το, με το Brexit. Ε, τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την πρόσβαση σε έγγραφα. Πέντε τα έχουμε διεκπαιρεώσει, δύο ακόμα εκκρεμούν. Έχω τονίσει και με τους συναδέλφους μου ότι για περιπτώσεις τέτοιες πρόσβασης στην, στα έγγραφα η δυνατότητα να βρει κανείς έγγραφα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει εφόσον δεν μπορούν να το κάνουν αυτό στα κράτη-μέλη ε, του. Στι αρχέ του έτου έγραψα και επιστολή και στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο Γιούγκερ για να του ζητήσουν ένα το δυνατόν πιο ενεργή σε ό,τι αφορά την διαφάνεια για τι ομιλίε Brexit. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτε να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για το πώ προχωρούν τα πράγματα, δεδομένου και τον δικτύπο που θα έχει τελικά. Ο Πρόεδρο Γιούγκερ ε, στην απάντησή του ότι θα υπάρξει μοναδικής, ε, μοναδικής ε, πρωτοφανής μάλλον ε, διαφάνεια αυτή τη φορά, κυρίως ό,τι αφορά τις, τα τελικά έγγραφα και τις τελικές οδηγίες. Δεν χρειάζεται να σας πω τι έχει γίνει από τότε. Όλοι βεβαίως περιμένουμε την σύνοδο του Δεκεμβρίου για να δούμε προς τα πού θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι κατά πάσα πιθανότητα, είναι πολύ, είναι πολύ πιθανό τα θέματα της διαφάνειας να μην λάβουν την προσοχή που τους αξίζει όταν περνούμε στα θέματα ε, εμπορικά κτλ. Συζητήσαμε σε μια σχετική διάσκεψη τα δικαιώματα των πολιτών. Το πεδίο βεβαίως, το τοπίο παραμένει ασαφές και βεβαίως Πάντα χρειαζόμαστε βοήθεια σε ό,τι αφορά την, τα δικαιώματα των πολιτών πριν και μετά τον Brexit. Οπότε όταν έχετε καλές ιδέε και προτάσει μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μαζί μα. Επίση, το κράτο δικαίου είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τη δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για κάποιου από του συναδέλφου ε, που ασχολούνται με χώρε όπου οι κίνδυνοι, υπονομ, ε, δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία. Πρόσφατα συναντήθηκα με τον κύριο Άνταμ Μπαλνέρ, τον Πολωνό ε, διαβασολαβητή και πραγματικά και ο ίδιος και η υπηρεσία του ε, εκτιμούν πολύ την ε, βοήθεια από τη δική μας υπηρεσία, από τη δική σας επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξεκολουθούν να ε, διατηρούν την ε, αρχή της, ε, του κράτους δικαίου σε όλες τις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η δουλειά μου έχει να κάνει κυρίως με τον κανονισμό 1049 του 2001 για, τη δημοσια... για την πρόσβαση στη δημοσία έγγραφα. Ως Επιτροπή υπεύθυνη για την νομοθεσία αυτή ξέρω ότι και εσάς σας ενοχλεί πάρα πολύ που έχει καθυστερήσει η αναθεώρηση από το 2011. Ξέρω ότι συμφωνούμε ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί για να καλύπτει όλους τις υπηρεσίες υπηρεσίε και τα θεσμικά όργανα και να τροποποιηθεί ώστε να, συμβα... να συμμορφώνεται με τι διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι ουσιώδου σημασία να ευρύνουμε το πεδίο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα θεσμικά όργανα που δεν καλύπτονται τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, α πούμε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακόμη και αν έχουν του δικού του κανόνε που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στα έγγραφα. Επίση, να πω ότι ο κανονισμό 1049 υπερισχύει οποιασδήποτε α, τεχνολογικής ε, εξέλιξης από το Twitter, το iPhone, δηλαδή τεχνολογία που χρησιμοποιούν ακόμα και οι έφηβοι τώρα και που δεν το μπορούσε κανείς να τη φανταστεί ότι θα υπήρχε στην, όταν γραφόταν ο κανονισμός. Ε, έχουμε ξεκινήσει μια δοκιμαστική φάση και μια διαδικασία fast track για την πρόσβαση σε έγγραφα και σε, και σε υποθέσεις. Πολλές φορές αν η γενική διαδικασία είναι πάρα πολύ μακροσκελή, ο ετών ε, σταματά, πάβει να ενδιαφέρεται πια να βρει το έγγραφο. Το άρθρο 15 της Συνθήκης Λισαβόνα επικεντρώνεται κυρίως στη διαφάνεια της νομοθετική διαδικασίας και υπό αυτό το πνεύμα, ε, φέτος ε, στις αρχές του έτους ξεκινήσαμε μια έρευνα για το πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και πώς συζητά την νομοθεσία στις Επιτροπές Κορεπέρ και στο Συμβούλιο. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τις γενικές πρακτικές της διοικητικές και Έχουμε έρθει και σε επαφή με τι υπηρεσίε του Συμβουλίου και κάναμε και μια δημόσια διαβούλευση πρόσφατα για να έχουμε τι απόψει και τη ε, Κοινωνία των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων. Και βεβαίω ευχαρίστω θα ακούσω τη γνώμη και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα στην ε, έρευνα αυτή του επόμενου μήνε. Η έρευνα ε, επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία, προσβασιμότητα και πληρότητα των εγγράφων του Συμβουλίου που βρίσκονται στο, στην ιστοσελίδα του ε, πρακτικές δημοσίευσεις ε, από τις διάφορες υπηρεσίες του ε, Συμβουλίου και επίσης διαφάνεια ό,τι αφορά τη θέση των κρατών μελών όπως λαμβάνεται αυτή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις, πολλές υποθέσεις καταλήγουν να μένουν στο Συμβούλιο χρόνια και βεβαίως οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνει η κυβέρνησή τους και τι θέση παίρνει. Το θέμα της διαφάνειας επίσης ε, μπορεί να ε, μειώσει την, ε, τον πειρασμό να λαμβάνονται όλες οι, αποφάσεις της Βρυξέλλες, εφόσον η ευθύνη βρίσκεται καμιά φορά και στα κράτη-μέλη. Τέλος, όπως ξέρετε, η υπηρεσία του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας ως κομμάτι ενός νέου, ε, νέου πακέτου για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Οπότε βεβαίω βεβαίως καλωσορίζουμε και εμείς την έκθεση ε, του 2017 που μελετά το πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει αυτό ως προτεραιότητα. Ξέρω βεβαίως ότι η έκθεση της Κομισιόν δεν κάνει καμία, κανένα, καμία αναφορά στο δικαίωμα της υποβολή ε, υποβολής καταγγελιών στον, είτε στο Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο είτε στον ε, διαμεσολαβητή ε, είτε στην πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτά είναι σημαντικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και όλοι μα πρέπει να τα προωθήσουμε μεταξύ όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω ότι αυτά θα ενταχθούν στην επόμενη έκθεση. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο πιέζει πολύ για να ενταχθούν και πάλι σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή σα σήμερα το πρωί, Πρόεδρε. Πολλά μας ε, είπατε κυρία Διαμεσολαβήτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλές πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα τα μέλη. Thank you to Mrs. O'Reilly for being here and your introduction. I would... ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγική σας ε, ομιλία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η Επιτροπή μας ε, θα έπρεπε να σας έχει εδώ πολύ πιο συχνά και εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα ε, όσα κάνετε για την διαφάνεια που πρέπει να έχουν και την πρόσβαση που πρέπει να έχουν οι πολίτες στα έγγραφα. Υπάρχουν τρεις υποθέσεις ενώπιον σας όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Επειδή σε μια έχετε ήδη πάρει απόφαση, θεωρήσατε ότι σε περίπτωση αιτήματο πρόσβασης ε, σε έγγραφα της ε, Κομισιόν και αν η Κομισιόν αρνηθεί να δώσει ε, έγγραφα, αυτό σημαίνει κακή διαχείριση, κακή διοίκηση. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου η Κομισιόν. Εδώ η Επιτροπή μας υποτίθεται ότι είναι διαρκώς ακούμε μάλλον ότι η Κομισιόν Λοιπόν θέλει να είναι θεματοφύλακας και θέλει να ε, απλουστεύει την νομοθεσία και τα λοιπά και να είναι προσβάσιμη και εδώ η άλλη άκρη πραγματικά και η άλλη όψη του νομίσματος ε, κακή διοίκηση και καμία πρόσβαση. Επίσης όσον αφορά τη διαδικασία fast track αυτές ε, είναι υποθέσεις, είναι διαδικασίες μάλλον οι οποίες τελικά παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και μέχρι να ληφθεί η απόφαση είτε από την υπηρεσία σας είτε από την Κομισιόν είτε το Συμβούλιο μέχρι να ληφθεί η απόφαση τέλος δεν έχει καμία σημασία, δεν, δεν έχει έννοια πλέον ε, και όσον αφορά την ε, απαιτήσει για ε, ασφάλιση μα όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν τώρα Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις επαφές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε, είχε με εκπροσώπους του εταιριών όσον αφορά την πρόταση για το PNR. Φαίνεται ότι η IBM μπορεί να έχει κάποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα αυτό και ότι το συζητούσαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ χρειαζόμαστε διαφάνεια γιατί πραγματικά αυτό μπορεί να επηρεάσει την εργασία μας. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι πολύ πιο ενεργό όσον αφορά αυτή την περίπτωση και να ε, ε, βοηθήσει να συνδράμει τον συνήγορο, την συνήγορο ε, του Ευρωπαίου πολίτη. Θα πρέπει να λογοδοτούν και το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Η πρόσκληση βεβαίως προς την ε, ε, Ευρωπαία ε, συνήγορο του πολίτη είναι σταθερή και διαρκής. Ναι, ναι, συμφωνώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, ότι θα πρέπει πραγματικά να είναι σταθερή και διαρκή η πρόσκληση. Η κυρία Αναγκόμες, ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Οραϊλή που ήρθατε. Συμφωνώ με την ε, Σοφή Ιντβέλτ ότι θα πρέπει να έρχεστε πιο συχνά γιατί η παρουσία σας είναι πολύ βοηθητική και μπορεί να γίνει ακόμα πιο βοηθητική στο μέλλον εάν τη χρησιμοποιήσουμε ακόμα καλύτερα. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πόροι. Πιστεύω ότι ιδιαίτερος Εν ώψη της λυπηρής ε, απόφασης της ε, Κομισιόν ε, να μην συνεχίσει την ε, ε, ε, πρόταση του Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την διαφθορά. Πιστεύω ότι στην ουσία αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματική λογοδοσία και απόδοση ευθυνών όσον αφορά την Κομισιόν και την βούλησή της για καταπολέμηση της διαφθοράς. Εδώ μιλάμε για το κράτος δικαίου, εδώ μιλάμε ε, για τον τρόπο ε, με τον οποίο ε, οι κυβερνήσεις μας, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, η Κομισιόν μπορεί να διαφαρεί από επιχειρηματίες και τα Ο ρόλος σας πάντα ε, υπήρξε πολύ σημαντικός και μπορεί να γίνει ακόμα πιο σημαντικός εν ώψη της έκθεσης που προετοιμάζει η ε, Κομισιόν ε, για τις λεγόμενες χρυσές θεωρήσεις, golden visas ή τις επενδυτικές διευκολύνσεις ας πούμε γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να δυναμητίζεται το σύστημα Σέγγεν και να δημιουργηθεί ανασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα που η Κομισιόν επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί με μια τέτοια έκθεση, πιστεύω ότι ε, θα ε, πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθούν και κάποια έγγραφα. Εγώ έχω δώσει πολλούς αγώνες έτσι ώστε ε, να μάθουμε τα ονόματα των ανθρώπων γιατί είναι περίπου 15.000 που έχουν επωφεληθεί από αυτές τις χρυσές βίζες, τις golden visas. Εμείς δεν ζητάμε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Ζητάμε μόνο τα ονόματά τους. Αυτό είναι ένα πεδίο ε, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, για όλους και εσείς μπορείτε να παρέμβετε σε αυτό. Τέλος, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Για την ε, Βουλγαρία. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Κομισιόν με χώρες οι οποίες δεν έχουν καλή διακυβέρνηση, όπως η Λιβύη. Έχουμε, ακούμε τρομερά πράγματα. Ακούσαμε ε, τρομερά πράγματα ε, για σκλαβοπάζαρα, για ε, σκλάβους, αλλά όχι μόνο η Κομισιόν και κάποια από τα κράτη-μέλη μας ε, καμώνονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι όλα γίνονται σύμφωνα με το κράτος δικαίου, ενώ έχουμε κατάφορες παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Ε, σε... γιατί Ξέρετε ότι το κράτος δικαίου προβλέπεται μέσω συγκεκριμένων κανόνων και όσον αφορά τις διακρατικές σχέσεις, ε, κυρίως όσον αφορά ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα προσφύγων. Αυτά ε, και σας ευχαριστώ. Η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ. Και εγώ μαζί με τους συναδέλφους μου θα σας ευχαριστήσω κύριε Ράιλι που βρίσκεστε ε, σήμερα εδώ και που ακούτε τόσο προσεκτικά ε, όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ε, που κάνουμε. Εγώ θα ασχοληθώ με τρία συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την μετανάστευση και την ανάγκη ε, μεγαλύτερης προστασίας ε, και αποτελεσματικότερης προστασίας ε, των προσφύγων είτε βρίσκονται σε διέλευση από την χώρα είτε διαμένουν στα κράτη-μέλη. Την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, το Συμβούλιο της ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ε, και σε σχέση και με την ενδοοικογενειακή βία σε σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στους μετανάστες στα κέντρα στα οποία διαμένουν ή κρατούνται. Επίσης, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και το ψήφισμα ε, το οποίο πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατάσταση στην ε, Μάλτα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω βάσει αυτού του ψηφίσματος να έρθετε σε επαφή και με τον συνήγορο του πολίτη της Μάλτας οι πολίτες της Μάλτας επανειλημμένα έχουν ε, ε, υποβάλει αιτήματα στον συνήγορο της Αμάλτας ε, για κακοδιαχείριση κτλ. Αλλά συνήθως η ερμηνείες του είναι πολύ ευρύς. Θα ήθελα επίσης για μία φορά ακόμα να σας ζητήσω να ε, ε, σκέψετε πάνω σε αυτό ε, που είπε και η Άννα Γκόμες για, γιατί εμείς δεν μιλάμε μόνο για θεωρήσεις ταξιδιωτικές βίζες αλλά μιλάμε για εθνικότητα δίνεται η υπηκότητα δηλαδή σε ανθρώπους περίπου ανεξέλεγκτα. Υπάρχει μια συμφωνία με την ε, ε, κυβέρνηση της ε, Μάλτας θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι διμερές ε, πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ε, μια χώρα δίνει υπηκότητα ε, σε κάποιον, αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται και άλλες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ποιος παίρνει την υπηκότητα, ποιο αντάλλαγμα έχει δώσει για να πάρει την υπηκότητα αυτή. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σε σχέση με το κατά εφόσον έχουν γίνει σεβαστές οι αρχές δικαίου. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και θα ήθελα να συγχαρώ ε, την ε, συνήγορο για τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζει τα θέματα. Αισθάνομαι ότι εδώ δίνουμε τον ίδιο αγώνα για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα. Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα και παρακαλώ να τα σκεφτείτε. Έχουμε τις συμφωνίες επανεισδοχής αλλά και τις άτυπες ρυθμίσεις επανεισδοχής

Είχαμε και χθε μάλιστα μια ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ε, τις επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής όπως ας πούμε αυτές που έχουμε με το Πακιστάν ε, να, δημιου... να αφήνονται λίγο στην άκρη ε, και να δημιουργούνται κάποιες άτυπες συμφωνίες. Ε, βλέπουμε ας πούμε την περίπτωση με το Αφγανιστάν, με την Τινησία, με την ακτή του Ελεφαντοστού, με πολλές χώρες της Αφρική, με τις οποίες δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη μετανάστευση ε, και με τον τρόπο αυτό καταπατείται το δικαίωμα ε, ελέγχου ε, από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε ε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επιστραφούν και όταν επιστραφούν τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς γιατί δεν, όταν δεν υπάρχει μια πραγματικά επίσημη συμφωνία δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν επιστραφεί, έχουν επιστρέψει συγγνώμη, στην χώρα τους ε, θα πρέπει να το, ε, να το δούμε το θέμα αυτό. Δεύτερο και τελευταίο, Πρόεδρε, το θέμα των μεταναστευτικών πολιτικών ε, που χρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μονάχα την ΛΥΜΠΕ ή μονάχα την Επιτροπή Ανάπτυξης. Είναι θέματα τα οποία είναι εγκάρσια υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αφορούν ε, τα Υπουργεία Εσωτερικών οποία, ε, και τα οποία αφορούν τη μετανάστευση και τα οποία χρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά το άρθρο 208 της συνθήκης λειτουργίας ε, ε, αναφέρει ότι ε, τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια αναφέρονται μονάχα στην καταπολέμηση της ένδυας. Εδώ χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτηθούν μεταναστευτικές πολιτικές και κινήσεις και πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να πάρουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα αυτά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πραγματικά θα εκτιμούσα εάν μπορούσατε να δείτε ε, αυτά τα ε, θέματα γιατί δεν υπάρχει ε, δημοκρατικός έλεγχος από τη δική μας πλευρά αλλά δεν υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος από την πλευρά της, υποδοχής, της χώρας ούτε από τη μία πλευρά δηλαδή αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά υπάρχει ανάμεξη στη διαδικασία. Okay. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε πώς συνεργάζεστε με τις διάφορες επιτροπές και τι γίνεται σε σχέση και με, την, με τον κανονισμό 1049 και την πρόσβαση στα έγγραφα και το ποιοι είναι οι, ποια, ποιος είναι ο λόγος για τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την πρόσβαση. Να επικεντρωθούμε λοιπόν εδώ σε αυτό ακριβώς. Βεβαίως τα καθήκοντά σας ε, αυξάνονται, διαφοροποιούνται, οπότε πείτε μας πώς βλέπετε με την συνεργασία με τις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Θέλετε να παραμείνει σε μια βάση ad hoc. Ε, η δική μας επιτροπή έχει ειδική ευθύνη για το θέμα της ε, πρόσβασης στα έγγραφα. Θέλετε να παραμείνουν έτσι σε μια βάση ad hoc τα πάντα και να είναι ευέλικτα, θέλετε κάτι πιο τυπικό, πείτε μας. Η απάντηση σε αυτό είναι θέλω αυτό που μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν μπορεί κανείς να δει τα έγγραφα, δεν μπορεί και να τα, να τα ερευνήσει, να τα ψάξει. Να απαντήσω καταρχάς στα ερωτήματα. Για την κυρία Νέτφελτ πρώτα. Νόμιζα ότι θα σας, ικανοποιεί, θα σας ικανοποιούσε η διαδικασία fast track. Ζητώ συγγνώμη για τις καθυστερήσεις βεβαίως που προέκυψαν και από δική μας ευθύνη. Και εμείς νιώθουμε την ίδια σύγχυση κάθε φορά που υπάρχουν ε, τέτοιες καθυστερήσεις και προβλήματα, κυρίως όταν δεν έχουμε πληροφορίες, όταν τις χρειαζόμαστε και κυρίως όταν χάνεται η σημασία και ο λόγος ύπαρξης αυτών των πληροφοριών. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Κάποιες από τις καθυστερήσεις οφείλονται σε προβλήματα από το δικό μου το γραφείο. Κάποιες έχουν να κάνουν και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ε, ε, θεσμικά όργανα, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή φτάσει κάποιος σε εμά. ας πούμε ότι είναι θέμα πρόσβαση τη Κομισιόν. Η Κομισιόν ήδη έχει δώσει την ε, απάντησή τη, είτε μέσω τη αρχική ε, διαδικασία, είτε μέσω τη διαδικασία προσφυγής. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ξαναγυρνάμε στην Κομισιόν και να τους δίνουμε μια παραπάνω περίοδο χρονική για να μας απαντήσουν και η απάντηση είναι ίδια με αυτή που παίρνατε στην αρχή. Οπότε Μιλάμε με την Κομισιόν, Έχουμε κάποιες ε, πρώτες επαφές, οι οποίες μάλλον φαίνεται να δουλεύουν καλύτερα πια. Και ελπίζω ότι τώρα που θα, από Γενάρη που θα ξεκινήσουν οι νέες διαδικασίες θα δείτε όντως τη διαφορά. Έχουμε και το θέμα αυτό των δύο εκκρεμών υποθέσεων σχετικά με το PNR με τις αιτήσει των κρατών μελών για συγχρηματοδότηση, αν θυμάμαι καλά. Η Κομισιόν διαφώνησε, ή τέλο πάντων εμείς διαφωνήσαμε με την ε, ερμηνεία της Κομισιόν ε, μιας απόφασης του δικαστηρίου για κάποιες διαδικασίες διαγωνισμών, οι οποίε εξισώθηκαν με την έτωση για συγχρηματοδότηση, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή και έτσι φαίνεται και η ανάγκη να τροποποιηθεί ο 1049 Και μάλιστα είπατε κι εσείς ε, κάτι παρόμοιο στη δεύτερη, στο δεύτερο σχολείο σας. Τι, όταν έγινε αντίστοιχο αίτημα από κάποιον πολίτη δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την, την επιχειρηματολογία. Το έπρεπε δηλαδή να ξαναξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Και αυτό είναι κρίμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κυρία Γκόμες. Ευχαρίστω να συζητήσουμε περαιτέρω για τα θέματα αυτά, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα θέματα που είναι αμυγός ε, αμυγού αρμοδιότητα κρατών μελών και τα υπόλοιπα που είναι αμυγθείς αρμοδιότητα. Οπότε, εμείς ευχαρίστως να έρθουμε σε επαφή μαζί σα για να το διερευνήσουμε. Σε σχέση με τη Μάλτα τώρα. Έχω πολύ καλές επαφές με τον Μαλτέζο συνήγορο του πολίτη Ο κύριος Πουλιτσίνο και ο κύριος ε, Μίψο ήταν οι προηγούμενοι ε, συνήγοροι. Έχουν ε, πραγματικά χαίρον μεγάλο σεβασμό στην, στη Μάλτα. Ξέρω ότι ο κύριος Πουλιτσίνο ήταν και πρόεδρος του δικαστικού σώματος. Νομίζω ότι και κάποιοι από τους προηγούμενους επίσης. Ευχαρίστω να συζητήσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά και το ψήφισμα. Ξέρω ότι η Μάλτα ήταν ε, στην πρώτη γραμμή την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για τις σχετικές συζητήσεις και βεβαίως αν μπορεί κάτι το γραφείο μου να κάνει, ευχαρίστως να το πράξουμε. Σε σχέση με τα αναπτυξιακά ταμεία, μου επέσανε προσοχή ατύπως το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ που το θίξατε. Και πάλι επανερχόμαστε σε αυτό που λέγατε εσείς κύριε Πρόεδρε για την πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό που μου είπαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι χωρίς να μπορούμε ακριβώς να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, που πάνε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε αν όντω χρησιμοποιούνται χρηστά ή όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθούν. Οπότε κάποιοι από τους συναδέλφους μου άρχισαν να ασχολούνται για να δουν ποια είναι τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα, ποια, αν δεν είναι διαθέσιμα γιατί δεν είναι. Είναι βεβαίως αρκετά διοικητική η δουλειά αυτή. Φυσικά είναι θέμα διαφάνειας έτσι ώστε να μπορούν και οι πολίτες αλλά και εσείς να αξιολογούν τα θέματα αυτά. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, σας ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι οι απαντήσεις που δίνετε υπονοούν ότι ερχόμαστε πιο κοντά και σε πιο επίσημο επίπεδο με την υπηρεσία σας εμείς ως Επιτροπή. Και βεβαίως η δουλειά που κάνετε προχωρά, γίνεται πιο λεπτομερής Μιλήσατε και για την διαδικασία fast track. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις βελτιώσεις και πραγματικά τις εκτιμούμε. Αλλά και στο μέλλον ας φροντίσουμε να έχουμε πιο στενή συνεργασία, πιο στενή σχέση. Μια που η αιτία τη συνεργασίας μας είναι ακριβώς η πρόσβαση στην πληροφορία και στα έγγραφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσία σα σήμερα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Uh, Να περάσουμε στο σημείο 11, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, για το, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Ασύλου. Συνάδελφοι, σημείο 11 λοιπόν, αν είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ε, θα έχουμε τώρα μια παρουσίαση της ε, ΕΑΣΟ, την παρουσίαση δηλαδή της ετησίας εκθέσεως της ΕΑΣΟ, όσον αφορά την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω λοιπόν στην Επιτροπή μας ε, τον εκτελεστικό διευθυντή, τον κύριο Χωσέ Καρέιρα. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η ετήσια έκθεση της ΕΑΣΟ περιλαμβάνει ε, ε, μια γενική θεώρηση όλων των εφαρμογών ε, ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσουμε και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και μια παρουσίαση διαφανειών ή βίντεο η ε, κατάσταση, η συλλογή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, ε, κατάσταση που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άσυλο και επομένως με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Καρέιρα ό,τι έχει να μας πει και μετά θα ακολουθήσει βεβαίως συζήτηση. Σας δίνω το λόγο κύριε Καρέιρα. I'm trying to find... Oh, uh, good morning. Good Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι παρό, παρούσες και παρόντες στο δωμάτιο. Θα ήθελα να σας πω ότι με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω εξ ονόματος της ΕΑΣΟ την ε, έκθεση που αφορά το 2016. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες, αλλά όχι και πάρα πολλές, γιατί ε, πραγματικά θα ήθελα κυρίως να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, να ακούσω εσάς δηλαδή περισσότερο. Ε, προς τα τέλη των διαφανειών θα δείτε και κάποιους πίνακε που αφορούν πληροφορίες για το 2017. Βρισκόμαστε ήδη στο Νοέμβριο. Ευελπιστώ ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί και η κατανόηση που δέχεται της κατάστασης. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις διαφάνειες. Πρώτη διαφάνεια λοιπόν είναι αυτή η οποία μας ε, δείχνει ε, του, του, τα, τις κύριες ε, διαδρομές που ακολουθήθηκαν το 2016. Έχουμε μια μικρή αύξηση 7% όσον αφορά τις αιτήσει. Πρέπει πρέπει ε, να ε, ξεκαθαρίσω ήδη ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στον αριθμό των παρατύπων ε, μεταναστών και την αύξηση των αιτήσεων στην ουσία. Η... δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο το 2015 είχαμε 1,4 ε, εκατομμύρια αιτήσει, το 2016 1,2 εκατομμύριο, σχεδόν 1,2 ε, και η μείωση είναι της τάξης του 7%. Πρέπει να σας πω κάτι που δεν βλέπετε, ότι έχουμε 600.000 ε, αιτήσει για την ώρα, δηλαδή περίπου το μισό από ό,τι την περσινή χρονιά. Οι κύριες χώρες υποδοχής το 2016 εξακολουθούν εξακολουθούν να είναι οι πέντε οι οποίες αναφέρονται στη διαφάνεια. Ε, ε, έχουμε την Γερμανία, την Ιταλία, την ε, Γαλλία, την Ελλάδα και την Αυστρία. Βεβαίως η πρώτη χώρα είναι η Ελλάδα και μετά κυρίως προωθούνται προς την Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία. ο αντίκτυπος αυτών των ε, εισόδων και μετά των αιτήσεων είναι ε, ο εξής. Ε, την προηγούμενη χρονιά, κυρίως ε, μετά από τον Απρίλη, η Ελλάδα και η Ιταλία κυρίως προσάρμοσαν την νομοθεσία, την νομοθεσία τους. Είδαμε ότι αυξήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις και περισσότερους χώρους το προσωπικό που ασχολείται με το άσυλο. Υπήρξε η οικοδόμηση ικανοτήτων μέσα από μοντέλα τα οποία ε, ε, υπήρχαν ήδη όσον αφορά ε, αστέγους ή όσον αφορά ιδιαίτερες κατηγορίες ανθρώπους. Η Ελλάδα και εν μέρη η Ιταλία άλλαξαν την νομοθεσία τους έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε πιο γρήγορες διαδικασίες ε, επίσης ε, και οι διαδικασίες ε, της νομολογίας και ενώπιον των δικαστηρίων έχουν διευκολυστεί. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση των προσφυγών γιατί όταν στις περισσότερες περιπτώσεις όταν οι αιτούντες λαμβάνουν αρνητική απάντηση προσφεύγουν για να συνεχίσουν την διαδικασία Βλέπουμε ε, γενικά ότι υπάρχει μεγάλη πίεση και ε, όσον αφορά την ε, στέγαση, όσον αφορά τις την αντιμετώπιση των πιο ευάλωτων ομάδων, όσον αφορά την, τις υποδομές υποδοχής κτλ. Βεβαίως εμείς δεν ασχολούμαστε με τις διαδικασίες υποδοχής, ωστόσο προσπαθούμε να παράσχουμε καταρτήσεις όσον αφορά την υποδοχή ε, όσον αφορά ε, την ε, κατάρτιση κυρίως των ατόμων που ασχολούνται με την υποδοχή. Νομίζω ότι ήδη τα είπα αυτά που δείχνει το, η διαφάνεια αυτή και να πω ότι εκτός από τις δύο ε, χώρες πρώτης ε, υποδοχής ε, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες συζητιούνται πολύ, υπάρχει ανταλλαγή απόψε όσον αφορά τις διαδικασίες συνεντεύξεων κτλ. Τώρα μιλάμε βέβαια ακόμα εδώ για το 2016 ε, που είχαμε 1,3 εκατομμύρια και παραπάνω ε, από αιτήσει. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, οι αιτήσει ε, καθυστερούν λίγο περισσότερο, παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο η μελέτη των αιτήσεων ε, γιατί υπήρχαν πριν αποφάσεις για ομάδες για τις οποίες η απόφαση ήταν εύκολο, εύκολη. Τώρα έχουμε λίγο διαφορετική εικόνα. Μετά από κάποια προβλήματα ε, ασφάλειας. Ε, αυτή τη στιγμή ε, οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν, μελετούν και θέματα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια και επομένως στην φάση της συνέντευξης προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν και το θέμα αυτό. Μεγάλος αριθμός αποφάσεων ε, έχουν ε, ληφθεί. Είχαμε αύξηση 34% ε, όσον αφορά τις αποφάσεις, τις πρωτόδικες αποφάσεις. Αυτός είναι πραγματικά ένας αριθμός ρεκόρ και οφείλεται και στις fast track διαδικασίες οι οποίες έχουν ληφθεί. Ε, γενική, ο γενικός λόγος ε, αναγνώρισης ε, επίσης έχει φτάσει στο 61% όσον αφορά τις πρωτόδικες αποφάσεις. Σε άλλες διαφάνειες που θα ακολουθήσουν θα δείτε ότι ότι πλέον προτιμούν την, την επικουρική ε, προστασία ε, παρά το καθεστώς ε, του πρόσφυγα γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές προστασίας τις οποίες είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε. Υπάρχουν οι απλές περιπτώσεις αιτήσεων ε, υπάρχουν περιπτώσεις επανένωσης ε, οικογενειών αλλά αυτό δυσκολεύει εάν ε, ο ετών δεν είναι ήδη πρόσφυγας. Έχουμε πολλές διαδικασίες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ε, περνούν από την ε, διαδικασία στην ανάγκη ε, ένταξης και ενσωμάτωσης. Εδώ γίνεται μεγάλη εστίαση. Ξεκίνησε η εστίαση αυτή το 2016 και συνεχίζεται και το 2017. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ένταξη, την προένταξη και στις πρώτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα και στις υπόλοιπες. Υπάρχουν επίσης χώρες χώρες ε, οι οποίες ε, ταυτόχρονα ε, αρχίζουν να αποσύρουν την προστασία όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τώρα, τα ποσοστά αναγνώρισης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δεν βλέπω εδώ τώρα τόσο μακριά, λέει ο μιλητής, αλλά θυμάμαι μερικά ότι απ' έξω η Γερμανία είναι λίγο πάνω από το 50%. Ε, για το καθεστώς των προσφύγων και ε, και έχουν επίσης και κάποιες άλλες μορφές αναγνώρισης. Η Ιταλία κάνει πολύ λίγα όσον αφορά ε, το καθεστώς του ε, ε, πρόσφυγα και πολύ περισσότερο όσον αφορά τα άλλα καθεστώτα. Στις περισσότερες χώρες βέβαια είναι το αντίθετο. Δίνουν το καθεστώς του πρόσφυγα πιο, σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Υπάρχει εδώ ένα στοιχείο σημαντικό που είναι το θέμα της εθνικότητας οι χώρες δεν έχουν όλες το ίδιο μείγμα εθνικοτήτων ε, μεταξύ των ε, προσφύγων ε, μεταναστών. Βεβαίως δεν εξηγεί αυτό από μόνο του ε, τις ε, διαφορετικές αποφάσεις και τα διαφορετικά ποσοστά. Ε, βεβαίως πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ερμηνεία που δίνεται για την κατάσταση, τον τρόπο προστασίας που μπορεί να πάρει η κάθε εθνικότητα κτλ. Μετά βεβαίως η υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσουν και να αναλύσουν ε, διεξοδικά τις υποθέσεις παρότι πίεζε ο χρόνος ε, υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες γιατί έχουμε ε, και ευάλωτες ομάδες, ανηλίκους διαφορετικά καθεστώτα προστασίας που οδηγεί και σε διαφορετικά προνόμια άλλα προνόμια δηλαδή έχει ο πρόσφυγας, άλλο αυτούς που χρήζει επικουρικής προστασίας. Και βέβαια και οι υπηρεσίε πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη. Είδαμε μια συγκέντρωση ε, δυναμικού υποδοχής. Κάποιες φορές ε, ήταν απαραίτητη ακόμα και συνεργασία με ΜΚΟ και με ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση των ευάλωτων ομάδων ε, ανάλογα με το κράτος μέλος, όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Και τα χώρε χώρες ε, ακολούθησαν το μοντέλο της ε, εδαφικής κατανομής. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουν περισσότερο και στο βορρά και στο νότο κατανομή σε όλη τη χώρα. Αλλά και η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν κατανείμει και τους ετούντες άσυλο και τους ε, πρόσφυγες ε, σε όλη την επικρατειά τους. Οι ανήλικοι πάντα αποτέλεσαν ε, σημείο ιδιαίτερης έμφασης σχεδόν το 1 τρίτο των ετούντων ήταν άτομα κάτω των 18, δεν σημαίνει ότι είχαν φτάσει μόνοι του. Υπάρχουν διάφορε διακρίσει μεταξύ του ανηλίκου και του ασυνόδευτου ανηλίκου. Δηλαδή, τα άτομα κάτω των 18 που έχουν φτάσει μόνο του στην Ευρώπη, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εδώ λοιπόν εξετάζουμε γενικά του ε, ανηλίκους κάτω των 18, του ετούντε έσυλο. Περισσότεροι είναι από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ, και το Πακιστάν, Νιγηρία, Ερυθρέα και Σομαλία. Δεν προκαλεί έκπληξη αυτό βέβαια. Επιβεβαιώνει την πραγματικότητα. Βέβαια, πολλοί από αυτούς συνοδεύονταν από μέλη της οικογένειάς τους, συνήθως τους γονείς τους, άλλες φορές από άλλους ε, συγγενείς. Κάποιες φορές υπήρξαν ε, και διαφωνίες για το κατά πόσο το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει την επιτροπή ε, του ανηλίκου ή όχι, εάν δεν συνοδεύεται από τους γονείς του. Τώρα, περνάμε στους ασυνόδευτους ανηλίκους, άτομα που έφτασαν στην Ευρώπη, άτομα κάτω των 18 και χωρίς συνοδό, μόνοι τους. Περίπου 65.000 ε, ετούντες είχαμε ασυνόδευτους ανηλίκους το 2016, 40% κάτω από το 2015, σημαντική μείωση. Παρά το και τα 65.000 υψηλό αριθμός είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 40% και λίγο παραπάνω ήταν από το Αφγανιστάν. Αυτό εξηγείται από ορισμένου κοινωνικούς παράγοντες που αναφέρουμε και στην έκθεση. Στα 5.000 λοιπόν, 40% από το Αφγανιστάν και 40% κάτω από το 2015. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Τώρα μέτρα προστασίας των ανηλίκων. Έχουμε εργαλεία για, την, ε, για τον καθορισμό της ε, ηλικίας, ε, την επιτροπή με τον όρο εργαλεία νοούμε υλικά για την ανείχνευση της ηλικία του ανηλίκου, αλλά και κατάρτιση οικοδόμηση δυναμικού για την ε, κατάρτιση των εργαζομένων που κάνουν τις συνεντεύξεις για να μπορούν να προσδιορίσουν την ε, ηλικία του ετούντος. Έχουμε κάνει πολλές ε, ειδικέ ενημερωτικέ εκστρατείε για τους ενηλίκους. Έχουμε παράσχει κατευθυντήριες γραμμές, έχουμε συνεργαστεί με τους ε, εργαζόμενους και με τους ανελίκους για να, τους, για να προστατεύσουμε τους ανελίκους κατά την άφηξή τους πρόσφατα. Συνεργαστήκαμε με τον ε, συνήγορο του πολίτη στην Ιταλία, γιατί εκεί το ποσοστό των ασυνόδευτων ενηλίκων είναι ιδιαίτερα υψηλό ακόμα και τώρα. για να τους δώσουμε τους τρόπους προσδιορισμού της ε, ηλικία, να διευκολύνουμε τη διαδικασία. αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από τον Αύγουστο. Προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε και να εργαστούμε και στα κέντρα υποδοχής για να ε, βοηθήσουμε τους ε, εργαζομένους προκειμένου και υποθέσεις ε, να αντιχάνουν επεξεργασίες πιο γρήγορα. Γενικά λοιπόν ο οργανισμός μας έχει εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση ε, του συντονισμού σε ό,τι φορά την ε, αντιμετώπιση και την επεξεργασία των αιτήσεων των ασυνόδευτων ενηλίκων. Περνώ τώρα στον Σεπτέμβριο 2017 και πάλι εδώ δεν βλέπω από τόσο μακριά την διαφάνεια. Να σας πω όμως ότι το 2015 είχαμε 1,4, 2016 1,3. Και τώρα έχουμε περίπου 600.000 ε, αιτήσει. Δεν είναι ακριβώς 50%, αλλά αν έχετε κατά νου ότι το 2017 είχαμε περίπου μισές από τις περσινές ε, αιτήσει, σχεδόν 50% πτώση έχουμε. Τώρα, οι επαναλαμβανόμενες αιτήσει. Δεν είναι κάτι απρόσμενο, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο όγκο δευτερογενών μετακινήσεων και διπλή καταμέτρηση στα σύνορα κάποιες φορές. Ετούντες που έχουν μετακατασταθεί και μετακαταθίσταται μετά και σε δεύτερο ή τρίτο κράτος μέλος. Μετά έχουμε 6-7%, 10% σε κάποιους μήνες Αυτό δείχνει ότι αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίε. Και μετά, μέσω του Δουβλίνου, επιτρέπουν ε, στο αρχικό κράτο μέλο ή μέσω των συμφωνιών με την κατάσταση σε πάνε στο επόμενο κράτο μέλο. Δεν λειτουργεί τέλεια αυτό το σύστημα, αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντε έχουν ε, οδηγήσει σε διπλή καταμέτρηση και σε διπλή υποβολή αιτήσεων κάποιε φορέ. Το θετικό είναι ότι το έχουν ανοιχνεύσει αυτό το πρόβλημα οι υπηρεσίες. Οπότε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εντοπίζεται η διπλή αίτηση και έτσι επεξεργάζονται μόνο την αρχική. Περνώ στην τελευταία διαφάνεια για την χώρα προέλευσης. Οι ίδιες είναι οι πέντε βασικές εθνικότητες, Συρία, Αφγανιστάν, Ιρακ, Νιγηρία και Πακιστάν. Τα πέντε κράτη-μέλη που ε, υποδέχονται τους περισσότερους έχουμε Ελλάδα και Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Μετά η πέμπτη άλλαξε. Δεν είναι πια η Αυστρία, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά Εν συντομία, για να σας παρουσιάσω αυτή την ε, πολύ διεξοδική έκθεση, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δώσατε το χρόνο. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Thank you very much and thanks for summarizing because we, I think we have quite a few questions. Colleagues, just keep... Ευχαριστούμε. Παρακαλώ στα δύο λεπτά. Γιατί στις 10.30 έχουμε επόμενο θέμα. Αναγκόμες παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε Κανένο για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας δείχνει ότι παρόλο το θόρυβο των κρατών μελών για να ε, δικαιολογήσουν ε, κάθε είδους μέτρα που λαμβάνουν, κυρίως επί της ασφάλειας, βλέπουμε ότι η εισρωή έχει ε, μειωθεί δραματικά το τελευταίο χρόνο. Να σας ρωτήσω λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα hotspot, τι γίνεται. Λειτουργούν ακόμα. Κατά καιρού ακούμε ε, ότι η κατάσταση σε κάποια από αυτά είναι δραματική. Ιδίως σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία ε, των ετούντων άσυλο να σας ρωτήσω επίσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου συμμετέχει σε οποιαδήποτε προγράμματα που αφορούν τη Λιβύη. Λιβύη. Και ποια είναι η γνώμη σας για τα τελευταία που βλέπουμε, τα γεγονότα που κάποιοι καταφτάνουν ε, στην Ισπανία. Και για τις εθνικότητες που αναφέρατε, νομίζω ότι πρόσφατα ε, και η Μαρακινή ήταν μεταξύ των χώρων αυτών, των εθνικότητων μάλλον. Τέλος. Μπορείτε να μας πείτε πώς τα κράτη-μέλη τα πάνε σε ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη αυτών των μεταναστών και προσφύγων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μέτσολα, παρακαλώ. Εγώ από πλευρά μου να σας ευχαριστήσω για τα όσα μας είπατε κύριε Καρέρα. Όταν μιλείτε μιλάτε για ανηλίκους. Μπορείτε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες. Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουν το καθεστώς ε, προστασίας οι ανήλικοι και τι συμβαίνει όταν δεν είναι επιλέξιμοι. Γιατί συνέχεια μας ρωτούν για αυτή τη νέα γενιά ανθρώπων που φτάνει στην Ευρώπη για να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον, από ποιες χώρες έρχονται, πού πηγαίνουν και στο πλαίσιο της ε, αναθεωρημένης ε, πρόταση του Δουβλίνου που έχουμε υιοθετήσει και πρέπει το Συμβούλιο να προχωρήσει, θα υπάρχει ένα σενάριο όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνε που δεν τι αναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Με του ανηλίκου πάντα Έχουμε διαφορετική πολιτική θέση. Όμως θέλω να μου πείτε περισσότερα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία που μας δώσατε. Την ηλικία τους, από πού έρχονται και τι συμβαίνει όταν λάβουν τον καθεστώς προστασία ή όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας της αίτησης. Πρόεδρος. Είναι μεγάλη διαφορά και μεταξύ των ε, συνοδευόμενων και συνόδευτων ανελίκων. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να είστε σύντομοι. Η Σιλβίκη Γκυγιόμ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, καθυστέρησα λίγο. Δεν άκουσα λοιπόν ε, την παρουσίασή σας. Σαφώς και θα διαβάσω το έγγραφό όμως με μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να μεταφέρετε μια εντύπωση σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση των ε, ε, μεταναστών. Έχουμε δει κάποια βίντεο πρόσφατα που παρουσιάζουν ένα σκλαβοπάζαρο ουσιαστικά στην Αφρική. Δεν ξέρω ότι υπήρξαν κινήσεις σε μιας γαλλικής ε, υπηρεσίας ασύλου που, έχει, είχε πάει εκεί ε, σε αποστολή. Υπάρχουν άλλες τέτοιες αποστολές. Μπορούν να αναλάβουν αυτές οι υπηρεσίες την προστασία αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων ή μπορούμε να τους ε, αναθέσουμε σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλες χώρες. Ευχαριστούμε, κυρία Σερζιντίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Μπορείτε όμως να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για τον ρόλο του ΕΑΖΟ τώρα στην Ελλάδα. Επισκέπτομαι τα νησιά. Έχω συναντηθεί και με ε, τους υπαλλήλους αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιος είναι ο επίσημος σας ρόλος εκεί. Δεν ξέρω αν ασχολείστε πλέον με πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στην εντολή σας. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το σύστημα. Και δεύτερον, για τις ε, δευτεροβάθμιες ε, αποφάσεις, τι είδους τάσεις διακρίνεται. γιατί βλέπω την νέα κυβέρνηση που θέλει να αφαιρέσει το δικαίωμα ε, παρουσίας δικηγόρου ε, στα, στις πρωτοβάθμιες αποφάσεις. Μπορεί αυτό να πάει και στις δευτεροβάθμιες ενδεχομένω. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τάση σε όλα τα κράτη-μέλη για τις δευτεροβάθμιες αποφάσεις και ποιος θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος Αντιμετώπιση του. Ευχαριστούμε, Μπριγκίτ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Από τις διαφάνειες διακρίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε δύο μεγάλες ομάδες ε, προσφύγων. Αυτούς που πραγματικά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, το βασανιστήρια, την πολιτική δίωξη, αλλά έχουμε και μετανάστε οικονομικού, ουσιαστικά που φεύγουν εξαιτία ε, τη φτώχεια και των κακών προοπτικών. Ένα ερώτημα λοιπόν από πλευρά μου. Εσείς ω μαζί και με τις εθνικέ αρχές μπορείτε να ενημερώσετε τα κράτη-μέλη για τις ε, πορείες ε, της μετανάστευσης και τις επιπτώσεις που προκύπτουν για να αντιμετωπίσουμε μάλλον τις αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Μετά κάτι που έλειπε από τις σας είναι οι πληροφορίες για τις ε, μεταφορές υπό το Δουβλίνο, που και πάλι είναι δυνατές πλέον ακόμα και προς την Ελλάδα. Και τρίτον, το πρόβλημα που συνεχίζεται με τα διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα. Δεν διακρίνεται από τις διαφάνειες γιατί υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Εξαιτία του αριθμού των αιτήσεων εξαιτία διαφορετικών ερμηνεών για το καθεστώς του πρόσφυγα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί στην Πολωνία μόνο Μαροκινοί εμφανίζονται, ε, το οποίο μπορεί να εξηγήσει, για παράδειγμα, ένα χαμηλό ποσοστό αναγνώριση, ενώ σε άλλε χώρε πάνε μόνο Σύριοι. Και έτσι έχουμε ψηλό ποσοστό. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια άλλη εξήγηση. Η κυρία Ντφέλτ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καρέρα για την παρουσίαση. Θα διαβάσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο. Θα περίμενε κανείς ότι και θα υπήρχε μία συνέντευξη τύπου των 28 ηγετών των κρατών μελών και να μας παρουσιάζουν ε, αυτά τα στοιχεία. Γιατί ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες δημιουργούν και προβλήματα ε, στις συζητήσεις ε, διαμόρφωσης ε, συνασπισμού, κυβέρνηση συνασπισμού. Είναι σαφές τώρα ότι υπάρχει μία πτωτική τάση, δεν αποτελεί πρόβλημα σε αυτό για το μέλλον, αλλά αν δούμε τα γεγονότα υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ αυτών των στοιχείων και των κραυγών αγωνίας ορισμένων πολιτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ επίσης στο θέμα των ε, ανηλίκων. Πρώτον, είχαμε ακούσει για 10.000 παιδιά που είχαν εξαφανιστεί. Δεν ήταν σαφές τελικά αν είχαν εξαφανιστεί, αν είχαν καταγραφεί. Μπορείτε να μας πείτε τελικά τι συνέβη. Και κατά πόσο ε, διερευνάτε η τύχη τους. Δεύτερον, πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα της ε, ανάθεσης ε, επιτρόπου. Ήταν της Europol το ζήτημα, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος, ο Πίτερ Νίδρε Μίλλερ, ε, εισηγητής για τον Ιάσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρέρα για την παρουσίασή σας. Πολύ σύντομα ένα ερώτημα ή μάλλον σχόλιο Μας δείξατε διάφορα γραφήματα και υπάρχει διαφορά μεταξύ Δύσης και Ανατολής στην Ευρώπη. Ε, οι χώρες του Βίσεγκρατ, της Βαλτικής, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν συμμετέχουν καθόλου στο σύστημα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πώς ο ΕΑΖΟ μπορεί να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, πώς έχει η κατάσταση των προσφύγων σε αυτές τις χώρες. Εγώ έχω πολύ αρνητικές εμπειρίες από τη χώρα μου, αλλά φαντάζομαι ότι η κατάσταση δεν διαφέρει και σε άλλες ε, χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής. Έχετε λοιπόν στοιχεία για την κατάσταση των προσφύγων σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Πίτερ. συμφωνώ πολύ με την κυρία Νιτφέλτ για την ε, σημασία αυτής της έκθεσης. Παρακαλώ, κύριε Καρέρα, να απαντήσετε. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Easy questions, uh, all of them. So let's try to, uh, try to give um, Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα σας τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ξεκινώ με το πρώτο. Τι συμβαίνει στα hotspot. Στην Ελλάδα εξακολουθούν να λειτουργούν τα hotspot με το ίδιο μοντέλο. Από τις 20 Μαρτίου, 20 Μαρτίου του 2016 αποκλειστικά σχεδόν λειτουργούν υπό τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Και αυτό που κάνει ο ΕΑΖΟ εκεί δεν αφορά όλο το σύνολο των εργασιών. Εμείς ε, ενημερώνουμε ακριβώς μετά την άφηξη, κάνουμε όλη την οικοδόμηση δυναμικού και αυτό το κάνουμε γιατί η σύνθεση του έργου αλλάζει συνεχώς. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η εμπειρογνώμονε των κρατών μελών. Ποτέ δεν έχουμε επαρκή αριθμό και αυτό το αντισταθμίζουμε ε, με την συμμετοχή του δικού μας προσωπικού, το οποίο αριθμός αυξάνεται. Οπότε, από τη μία εβδομάδα ε, στην άλλη και από τον ένα μήνα στον άλλον αλλάζουν ε, οι υπάλληλοι και το προσωπικό που έχουν διαθεσή μας, έτσι πρέπει να υπάρξει επανακατάρτιση. Συνεχίζουμε το έργο σε ευάλωτες ομάδες και ανελίκους αλλά δεν έρχομαστε εμεί σε απευθείας επαφή μαζί του. Αυτό είναι θέμα των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών υποδοχής στην Ελλάδα ειδικότερα. Στην Ιταλία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ειδική αρχή για τους ασυνόδευτους ανηλίκου, με τους οποίους εργαζόμαστε από τον Αύγουστο. Τα hotspot λοιπόν εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το ίδιο μοντέλο, ιδίως επειδή τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ε, ε, υπάρχει και πάλι αυξητική τάση στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ακόμα δεν μπορώ να σας βγάλω ένα μέσο όρο για τη χρονιά. Όμως υπήρξε σημαντική αύξηση. 5-5.500 το μήνα στην Ελλάδα οι αφήξεις στην Ιταλία πολύ λιγότερες. Αλλά και πάλι σημαντική η αύξηση. Αποτυχία για τη Λέσβο ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό έχουμε αποχωρήσει από τα hot spot. Ε, κρατάμε τις εγκαταστάσεις ε, εντός των hot spot, αλλά έχουμε δικά μας γραφεία και εκτός, το οποίο ουσιαστικά διπλασιάζει το δυναμικό μας. Είναι και θέμα ασφάλειας και πολλά κρατημέλη το έχουν ζητήσει. Οπότε για τα hot spot γενικά δουλεύουμε τον ίδιο τρόπο όπως πέρυσι, όπως μέχρι τώρα. Δεν μπορώ ακόμα να προβλέψω ότι θα συμβεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουμε έτσι και το 2018. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου για τη Λιβύη. Δεν ε, ε, έχουμε εμπλακεί ε, στο σχέδιο υλοποίησης της Μάλτας, όμως Έχουμε ε, συμφωνήσει, έχουμε υπογράψει τη συμφωνία για την επιχείρηση Σοφία, όπου δίνουμε μια light κατάρτιση ε, στους υπαλλήλου και στους ε, στρατιώτες όταν έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες. Τι ερωτήσεις να κάνουν, πρόσβαση σε διαδικασίες, δικαιώματα και να τους ενημερώνουν διαδικασία για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι να περιμένουν. Αυτή είναι η μοναδική μας συμμετοχή σε οτιδήποτε που ενδεχομένως να σχετίζεται με τη Λιβύη. Ε, τώρα, οι αφήξει ε, στην Ισπανία. Κατά μέσο όρο 2.000 κάθε μήνα για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Δεν είναι δικά μας τα στοιχεία, προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Frontex. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλές εξηγήσει. Μία από αυτές, η πλέον αξιόπιστη, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές πιέσεις στη Λιβύη και έχουμε νέες ε, διαδρομές από την Αλγερία, από την Τινησία και πάλι δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά. Επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάποιοι από αυτούς ε, φτάνουν στη Νότια Ισπανία. Αλλά εμείς δεν συμμετέχουμε, ούτε μας έχει ζητήσει κανείς ε, προς το παρόν να ασχοληθούμε με την Ισπανία. Οπότε δεν προβλέπουμε καμία ε, παρουσία μας στην Ισπανία. Για την κυρία Μέτσολα, τι συμβαίνει στους ε, ανηλίκους που δεν ε, χρήζουν προστασία. Η πλειονότητά τους βέβαια παίρνει το καθεστώς προστασίας, αλλά δεν έχω εδώ στοιχεία. Εάν δεν σας πειράζει, Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω γραπτός στο ερώτημα αυτό, γιατί χρήζει ιδιαίτερη προσοχής, είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή και ορθά. Θέλω να σας δώσω πλήρη απάντηση για την αντιμετώπιση των ε, ανηλίκων. Εμείς δεν συμμετέχουμε στα κέντρα υποδοχής ανηλίκων. συμμετέχουμε στην οικοδόμηση δυναμικού. Βοηθούμε τους υπαλλήλους ότι αφορά τον προσδιορισμό της ηλικία, τις ειδικέ ανάγκες. Προσπαθούμε ε, να συμμετέχουμε και να βοηθούμε, αλλά δεν μπορούμε προς το παρόν να παρεμβούμε. Αυτό θα προκύψει με τον νέο κανονισμό όταν εγκριθεί. Προτιμώ λοιπόν, αν δεν σας πειράζει, εντός ε, μιας εβδομάδας να σας δώσω μια πλήρη απάντηση που μπορείτε να δώσετε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας, για να σας δώσουμε ακριβή στοιχεία. για τον εισηγητή. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα. Α, η κυρία Γκυγιόμ. Ναι, δεν ξέρω αν ε, δεν το είπα καλά. Ξέρετε ότι υπάρχουν αποστολές που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, Γαλλική Υπηρεσία Ασύλου στον Ήγηρα και ε, προκειμένου άτομα τα οποία έχουν υποστεί βασανιστήρια ακόμα στο παρελθόν να ενταχθούν σε τέτοια ε, καθεστώτα προστασίας. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε τέτοια προγράμματα ή και ποια είναι η δική σας γνώμη. Και αν άλλες εθνικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ε, την ίδια αρχή διεθνούς προστασίας. Uh, ε, τα ξεκαθάρισα τα πράγματα. Ναι και όχι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο τέλος για να μην χάσω τη σειρά. Ο ρόλος του Άζος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ακόμα ε, συμμετέχουμε στην οριστικοποίηση του ε, προγράμματος ε, μετεγκατάστασης, έχουμε εκστρατείες ενημέρωσης, έχουμε ένα γραφείο αρρωγής, help Δεν κάνουμε την αξιολόγηση των φακέλων αυτό είναι θέμα των εθνικών αρχών και μετά για την μεταφορά στα κράτη-μέλη ούτε εκεί εμπλεκόμαστε. Είμαστε στη μονάδα Δουβλίνου στην Ελλάδα και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα το δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο μας ζήτησε να ε, διευκολύνουμε την ανάληψη των μεταφορών προς την Ελλάδα υπό το Δουβλίνο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Θα συζητηθεί και την επόμενη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε πώ μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι τι μεταφορέ Δουβλίνου προ την Ελλάδα. Ακόμα δεν γίνονται. Έχουμε κάποιου τέτοιου φακέλου, αλλά δεν συμβαίνουν ε, σε σχέση με τον αριθμό δηλαδή των πιθανών περιπτώσεων. Δεν έχουμε μεταφορέ. Ε, και υπό τη συμφωνία με την Τουρκία ε, έχουμε ρόλο. Τώρα, πώς μπορεί το δευτεροβάθμιο επίπεδο να είναι πιο αποτελεσματικό. Συνεργαζόμαστε και με τα δικαστήρια στην Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, με, τα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη. Βασικός πελάτης μας η Ελλάδα. Έχουμε πολλά πολλούς περιορισμούς, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς καταρτίζουμε τους δικαστές. Έχουμε υλικό λοιπόν ε, καθοδήγησης, κατάρτισης, ενημέρωσης ε, των δικαστηρίων και των εφετείων στην Ελλάδα. και διοικητική αροχή παρέχουμε προς τα δικαστήρια και τα φετία. Έχουμε λοιπόν υπαλλήλους που βοηθούν να προχωρήσει ο φάκελος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά με την ίδια την διαδικασία της έφεσης εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Νομίζω τα είπα όλα αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα. Το 2018 πρέπει να συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα, μην σας πω να αυξήσουμε την ε, συμμετοχή μας, γιατί υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, τα hotspot είναι γεμάτα όπως ξέρετε, η, η ταχύτητα επεξεργασίας ε, υπολείπεται του αριθμού των αφήξεων κάθε εβδομάδα, εδώ και πολύ καιρό. Οπότε θα είναι δύσκολη κατάσταση ε, και το 18. Βασικές αιτίες της μετανάστευσης και αντιμετώπιση τους. Να έχουμε τρεις πυλώνες της συνολικής μας ανταπόκρισης τα τελευταία τρία χρόνια. Στην αρχή είχαμε μπει σε ένα, ένα τρόπο διαχείρισης κρίσης με τα hotspot και το καθεξής. Μετά η Ένωση άρχισε να αντιμετωπίζει ε, τις ε, νόμιμες διόδους, τις βασικές αιτίες, τις χώρες προέλευσης, τους παράγοντες που οδηγούν σε, βασικές, ε, σε μαζικές ροές μετανάστευσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τον ΟΗΕ για του ε, μετανάστε και πρόσφυγες. Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται εκεί. Ήμουν πρόσφατα και στη Γενέβη. για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης ε, για το 2018. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο τομέα των εταιρικών σχέσεων. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Βασικές αιτίες λοιπόν, χώρες προέλευσης, χώρες διέλευσης, διαχείριση κρίσης. Πολλά έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του hotspot πλέον. αλλά υπάρχει και σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση και εμείς είμαστε τμήμα όλου αυτού. Θα έχουμε νέο φορέα σύντομα, υπάρχουν και νέες διαδικασίες σε υπό το πρόγραμμα επανακατάστασης, το οποίο θα αλλάξει σημαντικά το χάρτη. Εμείς ε, κλείνουμε το νομικό πακέτο. Στην Ευρώπη δηλαδή θεσπίζεται το, ο νέος οργανισμός ασύλου. Συνεχίσουμε, συνεχίζουμε να καταπολεμούμε τις ε, αιτίες της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο. Μας έχουν ζητήσει να αναλάβουμε ένα πιλωτικό έργο για τις ε, ιδιωτικές χορηγίες μετεγκατάστασης. και σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμα, αλλά έχουμε αρχίσει να, ασχολούμαστε με τις επαναγκαταστάσεις από την Τουρκία. Με τον Γενικό Διευθυντή διαχείριση μετανάστευσης της Τουρκίας για την οικοδόμηση ε, δυναμικού και την ενίσχυση του συστήματος ασύλου στην Τουρκία. Αυτό εν συντομία το έργο του ΕΑΖΟ για τις επιστροφές υπό το Δουβλίνο υπάρχει δίκτυο Δουβλίνου το οποίο αξιοποιούμε για τις επιστροφές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι περίπλοκη κατάσταση, ιδίω ε, με την Ελλάδα υπάρχει και διστακτικότητα σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης. Γιατί ουσιαστικά οι εθνικές αρχές ερμηνεύουν διαφορετικά την νομοθεσία, καθώς και η χώρα προέλευσης και τέλος έχουν διαφορετικές εθνικότητες που φτάνουν ε, στα σύνορά του Είναι διαφορετικά τα στοιχεία, λοιπόν, διαφορετική κατάσταση στι χώρες. Εμεί θέλουμε μεγαλύτερη σύγκληση. Ένα από τα καθήκοντα του νέου οργανισμού θα είναι η παρακολούθηση. Και σας διαβεβαιώ ότι το ποσοστό αναγνώριση σίγουρα θα παρακολουθείτε. Ο μελλοντικό οργανισμός λοιπόν ε, θα κατευθύνει και θα παρακολουθεί. Και ελπίζω έτσι ε, και σε καταστάσεις κρίσης να υπάρχει σύγκληση. Και έτσι να είναι μια ομοιόμορφη κατάσταση ό,τι φορά τα ποσοστά αναγνώρισης. Για τους ανηλίκους είπα ότι θα γράψω ένα δισέλιδο ε, σημείωμα όπου θα σας εξηγεί το έργο μας και με τα αντίστοιχα στοιχεία. Χώρες του Βίζεγκρατ και της Βαλτικής. Τι ισχύει εκεί. Πρόσφατα πήγα στην Πολωνία. Υπήρξε επιστολή της Πολωνίας προς τον ΕΑΖΟ για τα εθνικά ζητήματα, κυρίως έχουν από την Ουκρανία, Ρωσία και Γεωργία, κυρίως οικονομικοί μετανάστες και πολλοί από αυτούς ε, χρησιμοποιούν την Πολωνία ως ε, χώρα διέλευσης προς μια δεύτερη χώρα. Το γνωρίζουμε και έχουμε και ειδικά προγράμματα, αλλά δεν υπάρχουν, ε, δεν συμμετέχουμε στις διαδικασίες συνόρων, στις υποθέσεις, γιατί δεν είναι τόσο αυξημένοι οι αριθμοί. Οι εθνικές αρχές μπορούν ακόμα να τις αντιμετωπίσουν. Όμως παρέχουμε κατευθύνσεις και τους βοηθούμε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με την κυρία Γκυγιώμη Δημερός γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλετε από μένα, αλλά Έχουμε πολλά βίντεο, θα φέρω κάποια και στην επόμενη φορά, ιδίως στις υποθέσεις μας. Συνεργαζόμαστε με τη Γαλλία, κάνουμε εκστρατείες, ενημέρωσης για την Ιγυρία και άλλες χώρες. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Μπορεί να μην κατάλαβα το ερώτημά σας. Ε, ζητώ συγγνώμη. And, uh, once again... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Thank you, Mr. Um, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραϊρά. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να διαβάσετε την έκθεση αυτή. Είναι πραγματικά ουσιαστική σε ό,τι αφορά την ανάλυση των ε, πληροφοριών. Αναφερθήκατε ε, για το Δουβλίνο, για τις μεταφορές Δουβλίνου στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί το ρόλο αυτή και τα αποτελέσματά της είναι άλλη δουλειά. Είχαμε αρκετά δύσκολα ερωτήματα σήμερα για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το σύστημα ασύλου. Βεβαίω το υλικό που έχετε στα χέρια σας είναι ουσιώδες, δεν το συζητά αυτό κανείς. Και γι' αυτό θέσαμε τόσο δύσκολε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε και πραγματικά από τα στοιχεία που έχουμε είναι ε, πολύ σημαντικά αυτά που απορρέουν για το άσυλο, για τους μετανάστες κλπ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την παρουσίασή σας. Βεβαίως είναι ένα θέμα ανεξελίξη, αλλά σε αυτή τη φάση σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Και φυσικά θα ευχαριστούμε και τους συναδέλφους σας που δούλεψαν και μας παρέχατε όλη αυτή την ε, βιβλιογραφία. Και ευχαριστώ βεβαίως και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν. Προχωρούμε λοιπόν. Πάμε στο σημείο 12, συναδελφοί, σχέσεις με την Αφρική. Μετανάστευση και άσυλο και πάλι. I'll just pause while um, our colleagues come to the uh, podium. So colleagues, you may be aware that tomorrow we're going to have a high-level uh, conference on Africa. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σχέσεις με την Αφρική. Πολλά μέλη της Επιτροπής Λίμπερ είχαν ζητήσει να γίνει αυτή η διάσκεψη για την Αφρική για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα και σε σχέση με τα θέματα κλειδιά που μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή μας. Δεδομένου αυτού λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μια προπαρασκευαστική συζήτηση με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Θα μας παρουσιάσουν την κατάσταση σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής για τον τομέα της μετανάστευσης και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τις αντιπροσωπίες από τα διάφορα... Α, δεν είναι εδώ από τα διάφορα κοινοβούλια της Αφρικής. Θα φτάσουν, έρχονται. Ωραία. Άρα θα τους καλωσορίσουμε όταν έρχομαι. Έχουμε λοιπόν ε, μέλη της, ε, του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, της Εθνικής Συνέλευσης της Νιγηρίας και της ε, Συνέλευσης των Εκπροσώπων του Λαού της Τινησίας. Η συζήτηση σήμερα θα ασχοληθεί με, το, με την εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016 και, την, και τις αντίστοιχες εκθέσεις προόδρου και τις δήλωσεις της Βαλέτας του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2017 και, την, ε, και το καταπιστευματικό ταμείο ε, επιγούσε ανάγκη για την Αφρική. Ε, Βεβαίω όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επικεντρωνόμαστε φυσικά στην Αφρική, γιατί οι περισσότερε από τι αφήξει προ την Ευρώπη έρχονται από την Αφρική, κυρίω από τη Λιβύη, με πολλέ ζωέ να χάνονται στη διάρκεια του ταξιδιού, άτομα που την χάνουν ε, ε, εκμετάλλευση από του εμπόρου αλλά πολλέ πολλές φορές φαίνεται σαν να μην γίνονται αρκετές προσπάθειες από την ευρωπαϊκή πλευρά μαζί με άλλους διεθνείς παίκτες βέβαια όπως το ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η Αραβική Λίγκα για να διαχειριστούμε καλύτερα την κρίση τη μεταναστευτική και την προσφυγική. Η τη αρμοστία του ΟΗΕ επίσης και του πρόσφυγε και πολλέ ε, ΚΟ ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό για να βοηθήσουν τι εκστρατείας έρευνας και διάσωσης. Χαίρομαι που είναι διάφοροι συναδελφοί εδώ που μπορούν να μοιραστούν μαζί μας τις ε, απόψεις τους. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα έχουμε την ευκαιρία, βλέπω έρχονται και οι συνάδελφοι από τα Αφρικανικά Κοινοβούλια. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση για το θέμα αυτό. Οπότε θα ξεκινήσουμε αμέσως. Σιλβένα... η κυρία Μπριγκίτα Μάρκουσεν, η ε, αναπληρώτρια διαχειριστική διευθύντρια για την Αφρική τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Θα ξεκινήσουμε με εσά. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Χαίρομαι που είμαστε εδώ ε, με την συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Home, γιατί πραγματικά συνεργαζόμαστε στενά για το θέμα της μετανάστευσης. Θα σας κάνω εγώ μια παρουσίαση για το πού βρισκόμαστε και θα σας παρουσιάσω τρία βασικά στοιχεία. Θα ξεκινήσω καταρχάς λέγοντας το εξή. Πρέπει να ξέρετε κάποιοι από εσάς τους πέντε πυλώνες της πολιτικής δήλωσης ε, από τη Βαλέτα και το σχετικό σχέδιο δράσης. Εγώ θέλω απλώς να το τονίσω αυτό, γιατί εξεκολουθεί να αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούμε. Μετά, προχωρούμε στο εταιρικό, στην εταιρική σχέση. Ξέρω ότι συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Home θα σας μιλήσει και γι' αυτό. Αλλά πραγματικά έχουμε πάρα πολύ δουλειά ως προς αυτό. Με αυτό και μόνο ασχολούμαστε. Δηλαδή με τις ε, ε προετοιμασίες για τη σύνοδο τη επόμενη εβδομάδα, 29 και 30 Νοεμβρίου όπου η μετανάστευση είναι ένα από τα σημεία προς συζήτηση. Οπότε θέλω να σας κάνω μια αρχική ενημέρωση για το που βρισκόμαστε και ε, βεβαίως να ακούσω και τις ερωτήσεις σας σχετικά. Τώρα, τι κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Αν ακούσετε την Φεντερίκα Μαγκερίνη, θα ακούσετε ότι μιλούμε για μια ε, συνολική προσέγγιση, ε, ισόρροπη, δουλεύουμε για τις, πάνω στις γεωργικές αιτίε, αιτίες, πάνω στην νόμιμη μετανάστευση, προστασία των μεταναστών, αντιμετώπιση των ε, εγκληματικών δικτύων και επιστροφές, επανεισδοχές. Αυτά είναι τα πέντε βασικά στοιχεία πάνω στα οποία δουλεύουμε. Όλα αυτά συμφωνήθηκαν στη Βαλέτα. Μετά, Έχουμε μεταφράσει όλες αυτές τις ε, θεωρίες σε ε, διμερείς πρακτικές συμφωνίες, δράσεις με χώρες της Αφρικής. Θα ξέρετε τις πέντε πρώτες που επελέγησαν, τέσσερις στη Δυτική Αφρική και μία στην Ανατολική. Στη Δυτική Αφρική δουλεύουμε με την Ιγυρία, εγώ μόλις επέστρεψα μία αποστελή, με τον Ήγυρα, με το Μαλί, με τη Σενεγάλη και με την Αιθιοπία. Βεβαίως ε, υπάρχουν και άλλες ε, χώρες που έχουν ε, χρησιμοποιήσει αυτή την προσέγγιση τις εταιρική σχέση, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι πέντε αυτοί οι πυλώνες για τους οποίους σας μίλησα μόλις πριν. Τώρα, για την Σύνοδο Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, σε ό,τι αφορά το διάλογο που έχουμε και τη δουλειά που κάνουμε με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Αυτό που βλέπουμε, κυρίως για την Σύνοδο, είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον υπηρετικό διάλογο. Αν δείτε, ας πούμε, την Βαλέτα, εκεί ε, συζητήθηκαν ε, οι ε, διαδικασίες του Ραμπάτ και του Χαρτούμ. Αν δούμε τώρα την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, θέλουν μια ευρύτερη συζήτηση για διάφορα θέματα. Ας πούμε, τη διασπορά, τα θέματα που έχει η Αφρική με την εσωτερική της μετανάστευση εντός της Υπήρου, δηλαδή μετακίνηση προς την Νότιο Αφρική. Ένα διαφορετικό είδος δηλαδή διαλόγου που θέλουμε να ενισχύσουμε και θέλουμε να αποτελέσει το αποτέλεσμα που θα απορρεύσει από αυτή τη σύνοδο με την Αφρικανική Ένωση. Εμείς ε, θέλουμε να δούμε θέματα και κινητικότητας και μετανάστευσης Θέλουμε δηλαδή να έχουμε και το θέμα της κινητικότητας ως ε, κομμάτι της συζήτησης, κοινωνικο-οικονομικά θέματα, θέματα ασφάλειας και κοινωνικά θέματα και για την Ευρώπη και για την Αφρική. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία. Από, αυτό είναι το σημείο κίνησή μας για την ε, Σύνοδο θέλουμε να έχουμε και κάποιες ε, ναυαρχίδες όπως τις λέμε, να έχουμε δηλαδή κάποια απτά ε, παραδοτέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κοινή ανακοίνωση που είχαμε κάνει τον Ιούνιο είχαμε πει ότι θέλουμε να δουλέψουμε ε, και για την εσωτερική στην Αφρική μετανάστευση και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εγκληματικά δίκτυα. Μετά η Αφρικανική Ένωση ήρθε σε επαφή μαζί μας το Σεπτέμβριο και μας είπαν εντάξει είναι τα δύο αυτά θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, αλλά εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε και αυτόν τον υπηρετικό διάλογο για την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Και εμεί είπαμε αν αυτή είναι η δική σας πρόταση, ευχαρίστως. Εμείς είμαστε ανοιχτοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση να το συζητήσουμε, να δουλέψουμε τα θέματα αυτά. Οπότε βλέπουμε αυτά τα έξι, αυτές τις έξι θεματικές ενότητες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις βεβαίως, είμαστε το μέσο αυτών. Οπότε τα θέματα ακόμα είναι ανοιχτά. Εμείς απλώς θέλουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε το, από πού ξεκινάμε εμείς εμπόριο ε, μεταναστών ε, μετά είναι ε, παράνομη μετανάστευση και επιστροφές επανεισδοχές, διεθνή προστασία, τρίτο σημείο, τέταρτο εμβάσματα και διασπορά. Έχουμε λοιπόν την ομάδα των ε, διαπραγματευτών που έχει πάει στην Αντισαμπέμπα και ε, δουλεύει μαζί με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολλά τα ερωτήματα. Πριν περάσουμε στα μέλη, η Σιλβένα Πέστα, η αναπληρώτρια τμήματάρχης από τη Γενική Διεύθυνση Home, θα πάρει το λόγο. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε και πάρα πολλά ερωτήματα. Ευχαριστώ, θα είμαι όντως σύντομη. Απλώς να προσθέσω κάποια στοιχεία σε αυτά που ήδη ακούσατε. Βεβαίως η μετανάστευση βρίσκεται ε, στα πρώτα θέματα της, του θεματολογίου και στις σχέσεις μας ε, με τους Αφρικανούς εταίρους. Στην διάσκεψη κορυφής της Βαλέτα το 2015 οι ηγέτες μας ε, ε, συμφωνήσανε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ε, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της των χωρών της Αφρικής. Στις διαδικασίες της Ραμπάτ και του Χαρτούμ επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία αυτά και τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου για τη μετανάστευση επί τη βάση προηγουμένων προσπαθειών ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το πλαίσιο εταιρική σχέσης και επ' αυτού ε, βασίζονται οι σχέσεις με τους εταίρους μας. Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία βασίζεται στη διαφάνεια, στη ελληνική, στον επιμερισμό ευθυνών και στην ε, συνολική ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ θετικά αποτελέσματα με εταίρους όπως είναι ο Νίγηρας ας πούμε και αποτελέσματα όσον αφορά το τράφικινγκ, όσον αφορά τις παράνομες ε, διακινήσεις. Ε, οι παράνομες ε, κινήσεις έχουν μειωθεί ειδικά σε ορισμένες ε, περιφέρειες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες περιοχές στις οποίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και ε, ακριβώς ε, εμείς βοηθούμε ε, τους εταίρους μας σε όλα τα επίπεδα να αντιμετωπίσουν τα αίτια της μετανάστευσης, να αντιμετωπίσουν τις παράτυπες αναχωρήσεις, διαδικασίες επανεισδοχής. Εκεί κάνουμε επίσης και εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να κατανοήσουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως θα ήθελαν να μεταναστεύσουν τους κινδύνου και βεβαίω να τους γνωστοποιήσουμε και ποιες είναι οι νόμιμες οδοί ε, μετανάστευση. Και όσον αφορά αυτήν την νόμιμη μετανάστευση, εμπλέκουμε και τις χώρες ε, μέλη ε, σε διαδικασίες τέτοιου είδους τέλη Σεπτεμβρίου μάλιστα, μάλλον πριν δύο εβδομάδες μάλλον, ε, ολοκληρώθηκε η έκθεση για την νόμιμη ε, μετανάστευση. Επίσης έχουμε και το καταπίστευμα για την Αφρική που έχει κινητοποιηθεί ε, και περιλαμβάνει περίπου 117 πρωτοβουλίες για 2 δις ευρώ. Ε, ασχολείται με θέματα όπως η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης, δημιουργία κοινωνικής ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας κτλ. Υπάρχουν και κάποια σημαντικά ε, ε, κάποιες σημαντικές ημερομηνίες, η διάσκεψη κορυφής βεβαίως. Μετά θα έχουμε μια συνάντηση senior officials για τη διαδικασία του Χαρτούμ και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της Βαλέτα τον επόμενο χρόνο. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε αυτά τα επιπλέον στοιχεία. Έχουμε, και πρέπει να σας το πω αυτό, και εκπρόσωπο από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και από την Εθνική Συνέλευση της ε, Νιγηρίας. Θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε το λόγο μετά. Όμως τώρα θα δώσω το λόγο αμέσως στα μέλη. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους με τη ε, σειρά που τον ζήτησαν η κυρία Κιέγκε. Δύο λεπτά παρακαλώ, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Η Ευρώπη και η Αφρική ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ε, συνδεδεμένες ε, μοίρες αλλά ε, υπάρχουν ε, κοινά διακυβεύματα και προκλήσεις ε, αλλά και προϋποθέσεις σωστές με την προϋπόθεση βέβαια ότι και ευκαιρίες συγγνώμη πολλές με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα γίνει μια καλή εταιρική σχέση η οποία θα είναι τύπου win-win. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στα ωραία λόγια και στις εκδηλώσεις. Θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε την ανάπτυξη ανάπτυξη πολιτικών, κοινωνικών και όχι μόνο οικονομικών ε, στόχων. Ε, τα στοιχεία αυτά ε, είναι οι διάφορες εκφάνσεις του ιδίου προβλήματος και θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν έτσι ώστε να προωθηθεί η δημοκρατία, η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά δε το τελευταίο θέμα, θα ήθελα να βάλουμε επιγόντως στην ημερήσια διάταξη και το θέμα της Λιβύης. Ξέρουμε αυτά που συμβαίνουν στην Λιβύη τώρα και πραγματικά είναι ντροπή. Ε, θα πρέπει να δραχθούμε τις ευκαιρία του διαλόγου με την Αφρική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ο διάλογος ε, ε, Αφρική και Ευρωπαϊκής Ένωση όσον αφορά την μετανάστευση θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα όχι μόνο ανθρώπων που έχουν πολλά προσόντα αλλά και ανθρώπους με μικρότερα προσόντα. μη λησμονούμε το δημογραφικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην παραμελούμε λοιπόν τις δυνατότητες δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει μια νεανική ήπειρος όπως η Αφρική. Ε, θα πρέπει η κινητικότητα και η μετανάστευση να βασίζονται ε, ε, σε την ασφάλεια και επομένως θα πρέπει να ανοίξουν ασφαλείς διάδρομοι μετανάστευσης. Δεν να ζητήσω να καταλάβουμε ότι οι δύο ήπειροι έχουν και κοινά συμφέροντα αλλά και κοινά προβληματισμούς. Θα πρέπει η δράση να βασίζονται στην αλληλεγγύη και στη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ Σεσίλια. Η κυρία Βερζιά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμμερίζομαι την ε, αισιοδοξία των δηλώσεων που μόλις ακούσαμε. Εγώ δεν διαπιστώνω να υπάρχει ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση. η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι εκεί που ε, πεθαίνουν οι περισσότεροι που βρίσκουν το θάνατο εν τέλει οι περισσότεροι μετανάστες μεταξύ αυτών ε, μεγάλος αριθμός των ε, θυμάτων δηλαδή προέρχονται από την Αφρικανική ε, Ήπειρο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θωρακιστεί όσο γίνεται περισσότερο απέναντι στις αφρικανικές χώρες. Ε, κάθε ε, μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάνω από 2 εκατομμύρια ε, έγγραφα διαμονής αλλά όχι προς τις αφρικανικές χώρες και εγώ το λέω και το ξαναλέω εάν δεν ανοίξουμε νόμιμα κανάλια, νόμιμες διαδρομές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τότε θα κάνουμε ε, λάθος κίνηση και θα εξακολουθήσουμε να μετράμε νεκρούς στην Μεσόγειο. Θα αφήσουμε την κατάσταση στα χέρια των λαθροκινητών και των ε, διακινητών. Όλες οι πολιτικές ε, που ακούμε στην ουσία έχουν σαν στόχο την παρεμπόδιση της αναχώρησης ε, των ε, μεταναστών από τις χώρες της Αφρικής ή να τους επιστρέψουμε στις χώρες αυτές ανεξαρτήτως τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Υπάρχουν 244 εκατομμύρια μετανάστες απανταχού της γης. Επ' αυτών μονάχα 35 εκατομμύρια είναι οι Αφρικανοί. Το 85% των μεταναστευτικών κινήσεων ε, αφορούν ενδοαφρικανικές μετακινήσεις. Δεν είμαστε εμείς η πρώτη τους επιλογή και πρέπει να πω ότι οι πολιτικές μας δεν είναι πολιτικές συνεργασίας και εταιρική σχέσης ή αντιμετώπισης των βαθέων αιτίων της μετανάστευσης. Το αντίθετο μάλιστα. Ε, ναι, λέμε τα χρήματα της διασποράς. Τα χρήματα της διασποράς ξεπερνούν κατά τρεις φορές, αυτά τα εμβάσματα δηλαδή, ξεπερνούν κατά τρεις φορές την επίσημη χρηματοδότηση. Μερικές χώρες μέλη μάλιστα προσπαθούν να εντάξουν τα χρήματα αυτά της ε, ε, διασποράς, διασποράς ε, σε την αναπτυξιακή βοήθεια. Μα ποιον κοροϊδεύουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά την κατάσταση στην Λιβύη. Οι εικόνες που, έδειξαν, που έδειξε το, το CNN και που πραγματικά προκαλούν την οργή όλου του κόσμου, μα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να τις ε, ανεχτούμε. Ε, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό ε, η, ο, ο, ο πρόεδρος της χώρας μου ε, χαιρότανε γιατί ε, από τον Νίγηρα θα ε, υποδεχόταν 25 μετανάστες. 25, αν είναι δυνατόν. Ε, και ξέρω ότι θέλει να μιλήσει και έχουμε εδώ εκπρόσωπο από την ε, Να πω λοιπόν ότι η Ισία έχει πάρει περίπου ένα εκατομμύριο έχει υποδεχτεί μετανάστες από την Λιβύη. Θα πρέπει να κάνουμε συμφωνία μια κινητικότητα ε, ε, σωστή με τις ε, χώρες αυτές και πραγματικά η οργή μου ξεχυλίζει κύριε Πρόεδρε. Okay, um, thank you. Uh, Joseph please. Danke. Uh, Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα έχω. Καταρχάς, η κατάσταση στην Ανατολική Αφρική. Το είπατε ατροφηγός τι σκέφτεστε να κάνετε ως προς αυτό. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αποσταθεροποίησης που μπορεί να έχει πραγματικά βαρύτατες συνέπειες. Και βεβαίω οι άνθρωποι, αν επιλέγουν από την Ανατολική Αφρική να μεταναστεύσουν στην Ιεμένη, όπου σοβεί ο πόλεμο, φανταστείτε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Αφρική. Και επίσης, μιλήσατε για τη διασπορά. Τι θα μπορούσε κανείς να κάνει ώστε η διασπορά να, συνε... να συμμετάσχει πιο ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τζόσεφ, η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγο περίοργο είναι να είμαστε σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής ε, πολιτικών ελευθεριών και, για να μιλούμε, και να μιλούμε με την ε, Γενική Διεύθυνση Home και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για τις γενισουργούς αιτίες της ε, μετανάστευσης. Εγώ είμαι από, έχω αναπτυξιακό υπόβαθρο και το θέμα είναι θέμα ισότητας ή ανισότητας, κάτι που είναι η βάση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Μάλιστα έχουμε και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η, πολιτική μας, η εξωτερική πολιτική δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αναπτυξιακή συνεργασία και τους στόχους τους που είναι η μακρόπνοη απάλληψη, εκρίζωση της φτώχειας. Τώρα έχουμε όλο και περισσότερα κονδύλια από την αναπτυξιακή βοήθεια που δαπανώνται τελικά για σκοπούς μετανάστευσης και αυτό είναι προβληματικό. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια έκθεση ε, από, το Think Tank Klingendal που ε, ε, χρηματοδοτείται από την Ολλανδική κυβέρνηση για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις στο Ήγηρα οι οποίες τελικά οδήγησαν σε πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Έχουμε όντως μειώσει τη δυνατότητα λαθρεμπορία ανθρώπων, αλλά έχουμε οδηγήσει τελικά στους ανθρώπους στο να χάνουν οι άνθρωποι τι δουλειέ τους και, και στον Ήγυρα και γενικώ στην περιοχή του Σαχέλ. Ξέρουμε φυσικά ότι η περιοχή εκεί δεν είναι σταθερή και ακριβώς επειδή θέλουμε και ταχεία λύση για να σταματήσουν οι άνθρωποι να φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε στοχεύσει μια χώρα η οποία τελικά δεν βλέπει ε, να φεύγουν οι δικοί της οι πολίτες. Είναι μια χώρα διαμετακόμισης, είναι χώρα που περνάνε άτομα από την ε, ε αρχιτή του Αλλά ο Νίγηρας είναι μια πολύ φτωχή χώρα που λαμβάνει με χαρά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πολιτική λοιπόν που ε, ασκούμε εμείς δεν έχει να κάνει με τους γενεσιουργούς αιτίας της μετανάστευσης δεν έχει να κάνει με το να μην θέλει κάποιος να φύγει από τη χώρα του πια. Είναι, αυτό που κάνουμε είναι απλώς να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα φτάσουν στην Ευρώπη. Και αυτό είναι αντίθετο με οτιδήποτε πρεσβεύουμε σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Η αντιμετώπιση των γενοσυργών αιτιών της ε, ε, μετανάστευσης φυσικά είναι σημαντικός ε, στόχος, αλλά πρέπει να τον διαχειριστούμε διαφορετικά. Και επίσης, η ε, σύνοδος την επόμενη εβδομάδα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την νεολαία, όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά αν πάμε εμείς με την εσωτερική μας την ατζέντα και το εσωτερικό μας το θεματολόγιο, προσπαθώντας να κάνουμε την άλλη πλευρά να υπογράψει μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε λιγότερη μετανάστευση προς την Ευρώπη, νομίζω ότι τελικά δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Και γι' αυτό, αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει πραγματικά. As that contribution illustrated, this is a complex είναι περίπλοκο το θέμα αυτό, όντω. Και ξέρω ότι τα σχόλιά σα είναι πάντα ουσιώδη, αλλά παρακαλώ θα ξαναζητήσω να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Η κυρία Σίπολ. Ευχαριστώ. Θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια συμπεράσματα. Μιλούμε για τις, σε κάποια ερωτήματα. Μιλούμε για τη συνεργασία με τι αφρικανικέ χώρε και την αντιμετώπιση των γενεσουργών αιτιών τη μετανάστευση. Τι θα πει αυτό στην πράξη. Γιατί ακούμε πολλά που λένε ότι δαπανώνται κονδύλια για συνοριακούς ελέγχους για να, αποφύγουμε, να αποφευθεί η αναχώρηση από τις χώρες αυτές. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ενός πλαισίου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη. Τι κάνουμε συγκεκριμένα και ποιοι είναι οι τομεί πάνω στου οποίου επικεντρωνόμαστε. Επίση, νόμιμη μετανάστευση. Μιλούμε για νόμιμου τρόπου για του πρόσφυγε, μιλάμε για επανεγκατάσταση, μιλούμε για μόνιμους, νόμιμους ε, δρόμους ε, για άτομα που ψάχνουν μια θέση εργασία, ας πούμε για την μπλε κάρτα και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε το μέτρο αυτό στου διάφορου τομεί και σε συνεργασία με τα διάφορα κράτη-μέλη. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η συνάδελφο Αργεντίνη. Αν όντω θέλουμε μακροπρόθεσμα και βιώσιμα να αντιμετωπίσουμε ε, τι γενεσιουργού αιτίε τη μετανάστευσης, νομίζω ότι έχουμε μια ειδική ευθύνη σε ό,τι αφορά τι αφρικανικέ χώρε. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχει συνεργασία με άλλε ε, γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν που δεν ασχολούνται μόνο με την ανάπτυξη. Γενικώ, οι συνολικέ πολιτικέ μα για την αλληλεία, για τη γεωργία, για την ενεργειακή πολιτική, για το εμπόριο. Τι γίνεται, υπάρχει κάποια κρίσιμη σκέψη να αλλάξει η πολιτική μα ω προ αυτό για να βελτιώσουμε το μέλλον και για τι Αφρικανικέ χώρε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Μπριγκίτε. Η κυρία Γκόμε. Well, σε ό,τι φορά τι γενεσιουργού αιτίε τη μετανάστευση, δεν είναι μόνο η φτώχεια και η ανισότητα, είναι και η καταστολή, η καταπίεση, το οποίο συνδέεται βέβαια και με τα προηγούμενα, αλλά είναι ένα από του ε, λόγου που φεύγουν ε, από χώρες που, ε, όπως η Θεοπία που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια. Η Αιθιοπία καταραίει και αν καταρρεύσει η Αιθιοπία, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα από αυτά που βλέπουμε σήμερα και είναι απίστευτος και απαράδεκτος ο τρόπος που ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική δράση ε, κάνουν ότι δεν βλέπουν τα όσα συμβαίνουν ε, στην Αιθιοπία, όπου έχουμε ένα καταπιεστικό καθεστώς και βλέπουμε ότι χιλιάδε φεύγουν από την Αιθιοπία και όλο και περισσότεροι θα φεύγουν αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως πάνε τώρα. Θέλουμε λοιπόν δίκαιο εμπόριο, βιώσιμη ανάπτυξη, αλληλεία Τίποτα από όλα αυτά όμως ε, δεν αποτελεί αντικείμενο συντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή οποιοδήποτε άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, διευκολύνεται τις ε, παράνομες ροές που εξηγούν εν μέρη την ε, καταπίεση και καταστολή την κλεπτοκρατία που επικρατεί σε κάποιες χώρες ε, της Αφρικής και φέρουν τεράστια ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ίδιο ισχύει και στη Λιβύη. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Λιβύη, ότι ε, υπάρχει δουλεία στην πράξη, τέτοιε πρακτικές εξακολουθούν να υφίστανται. Ξέρουμε ότι πληρώνουν μισθοφόρους να χτυπούν κόσμο στην Λιβύη και δεν υπάρχει καμία συνανεργασία. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε καταρτήσεις για τη διοίκηση, για την ε, ε, συνοριοφυλακή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στην πράξη στη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα δεν έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ δεν μιλώ κατά της ε, στρατιωτικής επέμβασης στη Λιβύη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς αποχώρησε από τη Λιβύη και τους άφησε να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Και μέχρι να καταλήξουμε σε μια πραγματική στρατηγική, το μόνο που θα κάνουμε είναι να τροφοδοτούμε τους διακινητές. Γιατί εάν δεν επενδύσουμε σε νόμιμες ε, οδούς ε, μετανάστευσης, τι κάνουμε, ουσιαστικά ενισχύουμε τη σκοτεινή αυτή βιομηχανία των διακινητών. Πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους ε, προσκεκλημένους μας. Η κυρία Βίνμπεργκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίπου 60 εκατομμύρια πρόσφυγες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και πολύ θα ήθελα να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε. Δείτε τη χώρα μου, τη Σουηδία. Ε, δίνουμε τόσα χρήματα στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά εξαιτία των υψηλών επιπέδων μετανάστευσης που είχαμε προς τη Σουηδία τα τελευταία χρόνια, αναγκαστήκαμε να μειώσουμε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν βλέπουμε τόσους ε, ανθρώπους να ζουν σε προσφυγικούς ε, καταβλισμούς, το νόημα είναι ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε εκεί που βρίσκονται, στην Αφρική. Εμείς ε, στη Σουηδία αποφασίσαμε να υποδεχθούμε περισσότερους ε, πρόσφυγες και αυτό είναι καλός τρόπος να τους βοηθήσουμε ε, τους πρόσφυγες, αλλά αυτό ανεπόκειται στα κάτι μένει να το αποφασίσουν. Ή έτσι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Μιλούμε για τους λόγους της μετανάστευσης. οι πραγματικοί πρόσφυγες πολύ συχνά δεν καταφέρουν να βρουν θέση στην Ευρώπη. Πάνω από το 3% των μεταναστών, Μόλι 3% μάλλον των μεταναστών που έφτασαν στην Ιταλία ήταν πρόσφυγες, οι υπόλοιποι ήταν οικονομικοί μετανάστες. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πιο στοχευμένα το τι κάνουμε. Θα έπρεπε να έχουμε νόμιμες διόδους και νόμιμους διάβλους μετανάστευσης ε, να υπάρχει ποσόστοση αναγνώρισης ε, των ε, προσφύγων και να τους υποδεχόμαστε αυτούς. Αλλά όλοι όσοι έρχονται στην Ευρώπη δεν ξέρω με ποιο μοντέλο μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ η κυρία Νιτφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για την εισαγωγή τους. Εγώ συμφωνώ με, τις, με την κριτική και, τη, και τον προβληματισμό που έχουν εκφράσει οι συνάδελφοί μου. Πολύ ωραία μας ε, τα παρουσιάζετε ε, σαν ε, μία πολύ ωραία αναπτυξιακή βοήθεια. Ουσιαστικά τι πρόκειται για δωροδοκία των Αφρικανικών αρχών για να κρατούν τους μετανάστες εκεί. Αυτό είναι στην ουσία. Δεν πρέπει να ξεπλένουμε ούτε τους ηγέτες των Αφρικανικών αρχών από τις ε, ευθύνες τους, γιατί, όπως είπε και η Άννα Γκόμες, πολλές φορές ε, υπεύθυνοι είναι οι ηγέτες που στην καλύτερη περίπτωση είναι ανίκανοι, στη χειρότερη δικτάτορες. Ε, και είδαμε και πρόσφατα τον ηγέτη που προσπαθεί με νύχη και με δόντια να παραμείνει στην εξουσία στην ηλικία των 93 ετών, δηλαδή έλεος. Δεν ισχύει ότι αν δώσουμε πόρους σε κατασταλτικά καθεστώτα και δίνουμε και χρήματα ε, για τις, ε, για τους, ε, για τις δεν διευκολύνουμε τους ηγέτες αυτούς, τους δικτάτορες να συνεχίσουν την παρουσία τους στην εξουσία, την παραμονή τους. Και έτσι δεν δημιουργούμε προσφυγικές ροές. Μία άλλη μελέτη δείχνει ότι όσο αναπτύσσονται οι αφρικανικές χώρες και όσο ανεβαίνει το βιτικό επίπεδο, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητές τους να μεταναστεύσουν. Ποια είναι η γνώμη σας. Μετά, μιλήσαμε και για το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, δύο δις. Ε, δεν πρέπει να επενδύουμε στην Αφρική για να μην έρχονται Αφρικανοί εδώ, αλλά γιατί υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό έχει ανακαλύψει η Κίνα και επενδύει στην Αφρική δεν πρέπει να λέμε «Α, ας τους δώσουμε μερικά ψίχουλα για να μην έχουμε μετανάστευση». Θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική στρατηγική οικονομική συνεργασία με την Αφρική. Και τέλος, μια έκκληση προς εμάς περισσότερο, πρέπει να επαγρυπνούμε για να χρησιμοποιούμε τις δικές μας αρμοδιότητες ελέγχου του προπολογισμού. Γιατί πάντα εμείς ε, διαμαρτυρόμαστε για την ε, κακοδιαχείριση ε, των πόρων και την κακή εκτέλεση του προπολογισμού, όμως τελικά δεν κάνουμε και πολλά ε, εκ των προτέρων για να ελέγξουμε τον προπολογισμό. Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο και στις δύο μιλήτες για να απαντήσουν. Αλλά σας είχα προειδοποιήσει ότι θα είναι πολλά τα σημεία. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι μία συστηματική και σταδιακή αύξηση του έργου μας για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και αυτό θα οδηγήσει σε πολιτικές εντάσεις και σε άλλα ζητήματα όπως ανέφερε η κυρία Σαρτζεντίνη. Το δικό μου ερώτημα είναι η υπηρεσία εξωτερικές δράσεις πώς ε, το διαχειρίζεται όλο αυτό. Το είδαμε και στην Ελλάδα και αλλού. Στην Αφρική όμως τα προβλήματα είναι πιο βαθιά. Εμάς μας ενδιαφέρουν ε, ζητήματα κυρίως όπως είναι ε, η φύλαξη των συνόρων. Και πώς ε, εξασφαλίζεται η πολιτική λογοδοσία. Σε έναν βαθμό γι' αυτό είστε και εσείς εδώ σήμερα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τομέα αυτόν και ήθελα να το επισημάνω γιατί αυτό σίγουρα θα απασχολεί στην Επιτροπή και στο μέλλον. Ε, η προσεκλημένη μας, Πίνα Σάντσες, από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά παίρνω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ε, Επιτροπή σας. Βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να πω το εξή. Το θέμα της υποχρεωτικής μετανάστευσης είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο ε, και κατανοώ ότι είναι λόγος ανησυχίας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που ακούστηκαν εδώ κυρίως δε ε, με τους ε, βουλευτές που αναφέρθηκαν στα αίτια της μετανάστευσης, τις αιτίες δηλαδή που υποχρεώνουν τον κόσμο να μεταναστεύσει. Μία από τις αιτίες ε, στην Αφρικανική Ήπειρο είναι η ελλείψη της διακυβέρνησης, η πολιτική αστάθεια, η οποία ε, σπρώχνει τους ε, ε, νέους Αφρικανούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί βάσει σε βάθος διαλόγου, σοβαρού διαλόγου, διότι εν ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρος όπως και η Αφρικανική Ήπειρος στην ουσία είναι θύματα αυτών των πολιτικών ή των ελήψεων ε, στη διακυβέρνηση των χωρών της Αφρικανικής Ήπειρου. Αυτοί που εγκαταλείπουν την Αφρική το κάνουν για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Και Επομένως θα πρέπει να στηριχτεί ε, η Αφρική από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πραγματικά ε, ε, έχει μεγάλα προβλήματα λόγω αυτής της μάστιγας της μετανάστευσης. Το μέλλον μας είναι κοινό και θα πρέπει να είναι κοινέ και οι λύσεις. Η διάσκεψη ζωή της Αμπίτζα που δεν αφιερώνεται σε αυτό το θέμα όπως υπόθηκε και προηγουμένως θα μας δώσει παρόλα την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα το οποίο προβληματίζει την Ευρώπη και προβληματίζει και την Αφρική. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι για μία ακόμα φορά η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτήν την ηθική υποχρέωση. Είναι ε, πολιτισμού, είναι ήπειρος σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επομένως θα πρέπει να βοηθήσει την Αφρικανική Ένωση και γενικότερα την Αφρική έτσι ώστε να βελτιώσει τις ε, διακυβερνητικές διαρθρώσεις της θα πρέπει να σταματήσει πλέον αυτή η απάνθρωπη κατάσταση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τζόνσον Ογκούμα από την Εθνική Συνέλευση της Νιγήριας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Ήρθα από την Νιγηρία για να σας ε, μεταφέρω ένα μήνυμα. Να σας πω γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι από την Αφρική. Οποτεδήποτε οι άνθρωποι ε, σε όλη την ιστορία τους. Δεν αισθάνονται άνετα σε ένα φυσικό ε, περιβάλλον, ε, μετακινούνται. Αυτό γίνεται και τώρα. Το ζήτημα βέβαια περιπλέκεται λόγω της διαφθοράς στην Αφρικανική Ήπειρο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ε, ηγεσία στις χώρες της ε, ε, Αφρικανικής Υπήρου, αλλά μεγάλο ποσοστό ευθύνης βαρύνει και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα, τα παρανόμως κτηθέντα των Αφρικανικών ηγετών βρίσκονται σε τράπεζες, βρίσκονται σε άλλες υπήρους. Φεύγουν οι άνθρωποι από την Αφρική λόγω ε, του λοιμού, λόγω του πολέμου, λόγω της ε, διαφθοράς. Όταν ε, ήρθατε εσείς στην Αφρικανική Ήπειρο εμείς δεν σας διώξαμε. Ε, πήρατε ένα μέρος των πρώτων υλών. Ε, πήρατε ένα μέρος της ε, οικονομίας. Τότε η μετανάστευση δεν ήταν κακή. Ενώ τώρα βλέπουμε τα χρήματα των διαφθαρμένων ηγετών να επενδύονται αλλού. Εμείς σαν Αφρικανοί είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε ε, στην ε, Ήπειρό μας. Θα πρέπει να διώξουμε αυτούς τους ηγέτες. Βοηθήστε μας να το κάνουμε. Βοηθήστε μας ε, όταν αυτοί οι άνθρωποι κλέβουν ένα μέρος του πλούτου μας. βοηθήστε μας να τους διώξουμε. Ε, κοιτάξτε, και στο Ελσίνκι ε, εσείς όταν έρχομαι ε, ε, ή οπουδήποτε αλλού, εσείς αποφασίζετε τι θα κάνετε με μένα, τι θα πληρώσετε για μένα, με ποιο τρόπο θα με απασχολήσετε. Αυτό δεν είναι δίκαιο θα πρέπει δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, να ξαναδείτε λίγο, να αναθεωρήσετε τις ε, πολιτικές σας. Οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα ε, να ζουν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, σε ένα δίκαιο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον χωρίς πόλεμο. Ζητώ συγγνώμη, ε, θα ξαναμιλήσετε και αύριο. Δυστυχώς, λέει ο Πρόεδρος, δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε χρόνο. Ε, εσείς θίξατε πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Καλήφα από την συνέλευση εκπροσώπων του λαού της Τινησίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήρθαμε από την, την Ισία για να σας μεταφέρουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα. Η εταιρική σχέση με την Ευρώπη είναι θεμελιώδου σημασίας για την Αφρική. Ε, αφορά θέματα ασφάλειας, εμπορίου, ε, ανάπτυξης οικονομικής και κοινωνικής ε, και μετανάστευσης ε, και ε, όλα αυτά ε, από την οπτική γωνία της νεολαίας που θα αποτελέσει και κύριο στοιχείο της συζήτησης. Το θέμα αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Αφρικανική Ήπειρο. Πώς μπορούν να λυθούν τα ζητήματα κατάρτισης και απασχόλησης. Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία τους οδηγούν στη μετανάστευση. Είναι σημαντικό σημαντικό να μιλήσουμε και για διμερεί συμφέροντα προς όφελος των καλών σχέσεων που προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει με την Αφρική. Πρέπει να περάσουμε πλέον σε μια πραγματική αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική καλή διακυβέρνησης. Η Αφρική πρώτα απ' όλα θα πρέπει σήμερα να εκφράζεται με μία φωνή για να αντιμετωπίσει με σωστό τρόπο τα προβλήματα. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα είναι πώς να μειωθούν οι ροές των νέων που είναι ασυγκράτητοι ε, όσον αφορά την έξοδό τους, όσον αφορά την φυγή τους από τις χώρες τους και που καταλήγουν σε πολλές περιπτώσεις σκλάβοι να πουλιούνται στα σκλαβοπάζαρα νότια της Τρίπολης ε, στην ε, Λιβύη η διάσκεψη Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καθορίσει κοινούς στόχους και κοινούς τρόπους αντιμετώπισης. Η διάσκεψη αυτή οφείλει να θέσει τους νέους στο κέντρο των συζητήσεων θα πρέπει να ε, προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες ε, θα υποβληθούν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ε, η Αφρική είναι η πιο νεανική ήπειρος σε όλο τον κόσμο. Η δομή ο, ο πληθυσμός της ε, ε, στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι κάτω των 20 ε, ετών. Θα πρέπει επομένω να δώσουμε στους νέους αυτού ανθρώπους τη θέση τους, να δώσουμε ελπίδα, γιατί αυτή άλλωστε είναι και η ελπίδα για το μέλλον των δύο υπήρων. Επίσης θα πρέπει να τους μάθουμε το καθαρό περιβάλλον, έτσι ώστε να γίνουν πρωταγωνιστέ, να πάρουν το μέλλον των χωρών του στα χέρια του. Thank you. Thank you very much if Ευχαριστώ. Ξέρω ότι όλοι θα παρέμβετε εκτενέστερα αύριο και οι συνάδελφοί μας ε, από την Επιτροπή θα είναι παρόντες. Οπότε τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στην ε, Αναπληρώτερη διευθύντρια της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. πραγματικά συζητήθηκαν ε, πολύ σημαντικά ζητήματα και βλέπουμε ότι έχουν αντίκτυπο και στα θέματα προπολογισμού, στις πολιτικές που θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε παρακαλώ αν μπορείτε επικεντρωθείτε σε αυτά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Τα σημείωσα όλα. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις τους, τους ε, επισκέπτες ε, μας από τα Αφρικανικά Κοινοβούλια. Εγώ ήμουν στην Ιγυρία την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, ε, επισκέφθηκα τη Γερουσία σας, επισκέφθηκα τον Πρόεδρο και οι απαντήσεις μου είναι χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες. Καταρχάς, να σχολιάσω για τα όσα είπατε για την ε, σύνοδο με την Αφρικανική Ένωση. Μετά, θέματα λογοδοσίας, πολιτικές και να απαντήσω και σε κάποια επιμέρους σχόλια για τις διάφορες χώρες που θίξατε. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν έντονα συναισθήματα για τους τομείς αυτούς και αυτό είναι καλό νομίζω. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Θα το δείτε και στις υπηρεσίες της Κομισιόν αυτό. Και για εμάς, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, πρέπει να πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Φυσικά δεν υπάρχει ούτε εύκολη απάντηση, ούτε εύκολη λύση. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα και το είπατε και εσείς η Σύνοδος Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης δεν είναι σύνοδος για τη μετανάστευση. Η μετανάστευση θα είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο θα συζητήσουμε. Εγώ απλώς επικεντρώθηκα σε αυτό επειδή σήμερα μιλούμε για τη μετανάστευση. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Σύνοδος είναι για την νεολαία. Θα συζητήσουμε τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασία, την ασφάλεια και την ειρήνη. Βεβαίω και το θέμα τη μετανάστευση, βεβαίω και θέματα διακυβέρνηση. Αυτά είναι θέματα ε, ευρεία πολιτική που θα συζητηθούν. Και για πρώτη φορά προσπαθήσαμε από κοινού με την Αφρικανική Ένωση να, έχουμε την, ε, να κάνουμε μια καινοτομία, να εμπλακεί και η νεολαία στην διαδικασία αυτή. Έγινε τον Οκτώβριο μια σύνοδος για την ε, ε, νεολαία στο Αμπιτζάν και ήμουν παρούσα εκεί η δήλωση ακριβώς ε, που βγήκε από την σύνοδο εκείνη τροφοδοτείται στη σύνοδο που έχουμε αύριο. Για το τι ακριβώς θέλουν οι νέοι. Θέλουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα οι νέοι. Θέλουν ίσα πρότυπα μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση για να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα από τη μία ήπειρο στην άλλη. Αν θέλουν να, θέλουν να μπορούν να ε, εκλεγούν και να εκλέξουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία τα οποία βεβαίως μελετούμε. Υπάρχουν και ε, νέοι, μια ομάδα εδώ στην ε, στην, στις Βρυξέλλες, πήγανε στην Αμπιτζάν, στην Αντισαμπέμπα και θα μας δώσουν τις θέσεις τους. Αυτά για τη Σύνοδο. Μετά. Πού βρισκόμαστε εμείς στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση HOME, την DEFCO, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτά τα θέματα. Συμφωνώ με σας ότι αν δούμε τις γεννησιουργούς αιτίε. είπατε και εσείς ότι το μελετάτε και εσείς από την, πλευ... από την οπτική της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εμείς όμως στις εξωτερικές δράσεις κυρίως ασχολούμαστε με την κινητικότητα και τη μετανάστευση και για τη σύνοδο αύριο βλέπουμε και τη δυναμική του 90% της μετανάστευσης που συμβαίνει εντός της Αφρικανικής Ένωσης, ξέρουμε, της Αφρικανικής Υπήρου. Ξέρουμε ότι μόνο το 10% έρχεται προς την Ευρώπη και το ξέρετε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δυναμική και βεβαίως πρέπει να συνεργαστούμε με τους Αφρικανούς συναδέλφους και για τα θέματα που ισχύουν στην Αφρική. Για μας η μετανάστευση δεν είναι κατερνητικό. Είναι ένα μέρος της κινητικότητας, είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Βεβαίως, η λάθρο μετανάστευση, αυτή στην οποία αναφερθήκατε και εσείς και σχετίζεται με εγκληματικά δίκτυα, με λαθρεμπορία, ε, βεβαίως αυτό ενδιαφέρει και εμάς και εσάς να το αντιμετωπίσουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δημιουργούμε λοιπόν μια δυνατότητα για τα ταμεία και την χρήση των κονδυλίων. Αν δείτε το Ταμείο για την Αφρική, για τι επίγουσε ανάγκε, έχουν γίνει πολλές συζητήσει για το πώ θα δαπανηθούν τα κονδύλια αυτά, αλλά βλέπετε όλο και περισσότερο αυτά τα κονδύλια να πηγαίνουν στην ε, ενίσχυση των ε, υποδομών, των δυνατοτήτων διαχείριση, ε, των δυνατοτήτων επιστροφή των αφρικανικών χωρών αν δείτε πώς πάνονται τα κονδύλια, αυτή είναι η τάση που βλέπουμε και έχουμε αποφασίσει να προωθήσουμε. Τώρα, για τους συνοριακούς ελέγχους και τι κάνουμε. Αυτό σε καμία περίπτωση, ε, το έχει πει μάλιστα και είπατε εκπρόσωπος, η Ευρώπη δεν χτίζει τείχους, χτίζει γέφυρες. Είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία που θέλει να έχει συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους μου και με άλλους γείτονες. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω. Also border control. There is, for instance, the D5 Sahel. Έχουμε την μεικτή δύναμη για το Σαχέλ και που προέκυψε πάρα πολύ γρήγορα μια μονάδα που δραστηριοποιείται στην Πουρκίνα Φάσο, στο Μαλί, στον Νίγηρα, στη Μαυρετανία και το Τσάντ. Έχουν συνεργαστεί, οι ηγέτες των κρατών τους ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στις περιοχές μας. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία της περιοχής που ζούμε γιατί η κατάσταση χειροτερεύει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό να απαντούμε σε τέτοιες καταστάσει. καταστάσεις. Τρίτον, ξέρω ότι τελειώνει και ο χρόνος μου, αλλά κάποια από τα θέματα που θίξατε σε σχέση με την κατάσταση αναχώρα για τη Λιβύη, εχθές υπήρξε μια κοινή δήλωση μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης, του Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης και της ΥΠΑ της εκπροσώπου, την, της, ήρθε σε επαφή μαζί της το Σαββατοκύριακο για να συζητηθεί το θέμα της Λιβύης. Καταλήξανε λοιπόν σε μια πολύ σημαντική δήλωση όπου βεβαίως καταδικάζουμε στεναρά την κατάσταση και τα όσα γίνονται στη Λιβύη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή θέση. Εμένουμε σταθερά ε, στη συνεργασία μας και με τον ΟΗΕ και με άλλες, άλλους διεθνείς οργανισμούς για να προστατεύσουμε τα, τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στη Λιβύη και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Αιθιοπία. δεν θα πω ότι έχουμε στρατηγική εταιρική ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιθιοπίας. Προσπαθούμε όμως να δουλέψουμε πάνω σε διάφορα θέματα με την, με την Αιθιοπία, ακριβώς αναγνωρίζοντας το ρόλο που παίζει η χώρα αυτή στην Ανατολική Αφρική. Είπατε ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Αιθιοπία. Το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά επίσης γνωρίζουμε και τον οικονομικό και τον πολιτικό ρόλο που παίζει η Αιθιοπία. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή διάδραση, κυρίως και στα πλαίσια τη πολύ δύσκολη κατάσταση που επικράτησε πέρσι. Είναι πολύ στενό ο διαλογός μας, ευχαρίστως να τον ε, συνεχίσουμε για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δράσει αρκετά. Για την Ανατολική Αφρική δεν μιλήσατε βέβαια για συγκεκριμένε χώρες, αλλά Φαντάστηκα ότι θα μπορούσατε να αναφέρεστε στη Σομαλία και τον Νότιο Σουδάν. Δουλεύουμε πολύ στενά με την ε, ε, οργάνωση στην Ανατολική Αφρική για να δούμε πώς μπορούμε πολιτικά να λύσουμε την κατάσταση. Ε, Αν δείτε όμως τι συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν, Πραγματικά είναι τρομακτική η κατάσταση. Αυτά που υποφέρουν οι άνθρωποι στο Νότιο Σουδάν είναι τραγικά. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν. Και σίγουρα οι άνθρωποι που μετακινούνται στην περιοχή εκεί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Τη γνωρίζουμε λοιπόν την σοβαρότητα της κατάστασης και συμμεριζόμαστε ακριβώς τις ανησυχίες σας. Τέλος, το θέμα του Νίγηρα. τι γίνεται, αν όντω χάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους λοιπά, Μας ρωτήσατε. Έχω πάει αρκετέ φορές στον Ήγηρα. Και όταν μιλά κανείς με τις αρχές της χώρας, η αύξηση των ε, ε, διερχομένων από τον Ήγερ Είναι πραγματικά σημαντική και κάπως πρέπει αυτή η ροή να τύχει μιας διαχείρισης. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την πολιτική κατάσταση στον Ήγερα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση την πολιτική μεταξύ του Βορείου Νίγηρα και του τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ συνήθως στην γενική μας, από τη γενική μας διεύθυνση στην Αφρική είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η πολιτική μας ανάλυση να είναι σωστή για το κατά πόσο αντιμετωπίζουμε τη μετανάστευση σωστά και ποια είναι η κατάσταση της χώρας. Και μετά βλέπουμε και τη Γενική Διεύθυνση της ε, Home και τη Γενική Διεύθυνση DEFCO με τους εμπειρογνώμονές τους και πώς μπορούν και αυτοί να μας βοηθήσουν. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις διάφορες ε, χώρες, όλες αυτές που σας ανέφερα και προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους υπεύθυνου που μπορούν να βοηθήσουν ως προς αυτό. Σταματώ εδώ γιατί τα θέματα που θίξατε θα μπορούσαμε να τα συζητούμε μέχρι αύριο, οπότε καλύτερα είναι να τα συζητήσουμε όντως αύριο που θα είναι και η υπατή εκπρόσωπος παρούσα και να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο. Thank you. Ευχαριστώ. Μίλησατε για τις ζωές που χανόνται στη θάλασσα. Πράγματι, τα στοιχεία είναι σοκαριστικά. 2.750 φέτος. Όμως και πάλι είναι... υπάρχει μια πτώση σε σχέση με πέρσι, χάρη στις κοινές μας προσπάθειες. Και μπορούμε να αναφέρουμε και τους πάνω από 2.000 τις χιλιάδες ε, διασωθέντες από την Ιταλική ακτοφυλακή ε, και τους χιλιάδες που έχουν σωθεί στη θάλασσα από την ε, Λιβική ακτοφυλακή. Τώρα, αν οι νόμιμες δίωδοι αφορούν μόνο την επανακατάσταση, όχι, τη μετακατάσταση μάλλον όχι, Υπάρχουν κοινέ προσπάθειε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πιλωτικά προγράμματα σχετικά με την εργασιακή μετανάστευση, labor migration. Θα σα ενημερώσουμε, ελπίζουμε στο μέλλον. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και μαζί με τους εταίρους μας ανά τον κόσμο ε, εργαζόμαστε επί ενός παγκόσμιου ε, συμφώνου για τη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε και βλέπετε ότι ε, αυτό το θέμα δεν μπορεί να καλυφθεί στο περισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα έχετε και τη συνεδρίαση αύριο με ισχυρή εκπροσώπηση τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα τα πούμε λοιπόν και αύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπηρεσία Εξωτερική ε, Δράση και την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. και τους συναδέλφους για τα ερωτήματά του. Δεν θα σταματήσει εδώ αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, στις 11.30 ξεκινάει η συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν.